Uh, uh, uh, Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ να αρχίσουμε. Έχουμε λίγο καθυστερήσει. Ξέρω ότι ο Επίτροπος Μπορτζ ε, ήθελε να συναντήσει κάποιους από τους συναδέλφους. Χαίρομαι που είστε εδώ. Ξέρω ότι θέλετε να πάρετε και το λόγο. Οπότε θα ήθελα να ζητήσω τον Επίτροπο να είναι ε, συνοπτικός και παράλληλα να μας ενημερώσει. Για πρώτη φορά σας καλωσορίζουμε εδώ ως ε, ε, συμμέτοχος στο πλαίσιο του διαρθρωτικού διαλόγου. είναι επίσημο καθήκον σας, αλλά χαιρόμαστε όλος ιδιαίτερος που σας ε, έχουμε εδώ μαζί μας ε, για να μας πείτε ποιες θα, ποια θα είναι τα μελλοντικά σας σχέδια και ε, για την τρέχουσα κοινοβουλευτική θητεία, αλλά να μας πείτε και για διάφορα επιτεύγματα ενδεχομένως. Η Πάολα Τεστόρη είναι εδώ μαζί μας. Χαίρομαι όλος ιδιαίτερος. Σας καλωσορίζω. Το μόνο που μένει λοιπόν είναι να σας δώσω το λόγο, Επίτροπε μπόλτς. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, ε, βλέποντα τα τελευταία πέντε, ε, τις τελευταίες πέντε μήνες ε, όταν έλαβα το, ανέλαβα καθήκοντα στην ίδια και όλας αίθουσα, πρέπει να πω ότι έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο. Ε, χάρη στη συνεργασία με την Επιτροπή σας και σε γενικές γραμμές ε, με το Κοινοβούλιο για τα θέματα ε, των καταναλωτών. Αναμένω τώρα εναγωνίως στην έκθεση της ατζέντα για τους καταναλωτές που βασίζεται στην ασφάλεια, στην εκπαίδευση, την επιβολή και την εκπαίδευση, τους τέσσερις τους πυλώνες και την οποία προετοιμάζεται από ό,τι κατάλαβα θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια του Μαΐου. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εντατικοποιεί τις προσπάθειές της για να συνεχίσει τις ε, ε, πρωτοβουλίες της ατζέντα των καταναλωτών και ειδικότερα την ψηφιακή ατζέντα επαριθμών 2. Θα ήθελα να δώσω λίγο περισσότερε πληροφορίε για, τις τέσσερις, του τέσσερι αυτού πυλώνε. Καταρχά, την ασφάλεια. Νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει πολύ για το θέμα τη εποπτεία τη αγορά και τη ασφάλεια των προϊόντων ε, βάσει ε, τη έγκρισή μα ε, το Φεβρουάριο. Ε, κανονισμός, ε, για, νέος κανονισμός για την ασφάλεια των προϊόντων που εναρμονίζει κάποιους από τους κανόνες. Όπως γνωρίζετε ότι υπήρχε αυτή η διαφορά μεταξύ εναρμονισμένων και μη εναρμονισμένων προϊόντων. Κάποια ήταν αρμοδιότητα δική μου, κάποια του Επιτρόπου Ταγιάννη και προσπαθήσαμε κάπως να εξορθολογήσουμε τους κανόνες αυτούς ε, Υπάρχει επίσης και ένας νέος κανονισμός στο πακέτο για την εποπτεία της αγοράς. Θα υπάρξει μάλιστα και ένα σχέδιο εποπτείας για το 2013 με 2015 με 20 δράσεις ε, για να εξασφαλίσουμε ασφαλέστερα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας από τους στόχους μας λοιπόν είναι η χνηλασιμότητα των προϊόντων να είναι ευκολότερη, κάτι το οποίο βεβαίως θα ενθαρρύνει τη συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους μας ε, και ειδικότερα την Κίνα. Στο πλαίσιο αυτό, υποχρεωτική ένδειξη σε όλα τα καταναλωτικά προϊόντα προϊόντα της χώρας προέλευσης και άλλων στοιχείων αναγνώρισης των προϊόντων θα ε, αυξήσει τη γνώση της ε, αλυσίδας ε, προμήθειας. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και η Επιτροπή Πολιτισμού τώρα επιμένει στην ετικετοθεσία, για τη διαδικασία, για τη χώρα προέλευσης και ούτω καθεξής. Οπότε τουλάχιστον να ξεκινήσουμε με το ε, την ετικετοθεσία προϊόντων που δεν είναι διατροφικά. Ε, αν αυτό περάσει λοιπόν από το Συμβούλιο και από το Κοινοβούλιο θα σημαίνει πιο ε, καλή και πιο στοχοθετημένη επιβολή. Και επίσης βέβαια θα ενισχύσει και την εμπιστοσύνη στα προϊόντα που υπάρχουν στην ευρωπαϊκή αγορά. Παράλληλα ε, σκεφτόμαστε ποιες δράσεις μπορούμε να έχουμε για την καλύτερη ασφάλεια των υπηρεσιών. Μερικές φορές ξεχνούμε τις υπηρεσίες και κεντρωνόμαστε μόνο στα προϊόντα. Για το δεύτερο πυλώνα της ατζέντα, ε, τη γνώση των καταναλωτικών δικαιωμάτων, 15 ε, Μαρτίου ιδρύσαμε τον ιστότοπο που μπορούν να ανταλλάξουν ε, μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις, ε, ε, ενδιαφερόμενοι φορείς, διδάσκοντες και καταναλωτές. Υπάρχουν διαδραστικά εργαλεία για τη δημιουργία φόρα, για να υπάρχει πρακτική καθοδήγηση, 12 με, κυρίως προς άτομα 12 18 ετών, δεξιότητες καταναλωτών που όλοι χρειάζονται για την ενημέρωση των καταναλωτών έχουμε προβεί σε ένα πρώτο διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς, εκπροσώπους ε, οργανισμών καταναλωτών, ε, επιχειρήσεων και εθνικών αρχών για δύο βασικά ζητήματα. Πρώτον, ε, εργαλεία συγκρισιμότητας και δεύτερον, παραπλο, παραπλανητικά περιβαλλοντικές, παραπλανητικές αξιώσεις όταν κάποιο προϊόν παρουσιάζεται ως φιλικό προς το περιβάλλον, πράσινο ενώ δεν υπάρχει αποδεκτικό στοιχείο. Ε, Στη Σύνοδο για του καταναλωτέ 17 και 18 Μαρτίου ε, συζητήσαμε πώς είναι δυνατόν ε, και προσπαθήσαμε να δούμε πώς μπορούμε να ε, προχωρήσουμε. Η επιβολή της νομοθεσίας, ε, η διάσκεψη του περασμένου μήνα για τους καταναλωτές είχε αφιερωθεί στο συγκεκριμένο θέμα. Οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι ενώ η υπάρχουσα καταναλωτική νομοθεσία είναι αρκετά εκτενής, υπάρχει, υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερης αναμόνησης στην πράξη. Επομένως έγινε μια έκκληση κατά τη διάσκεψη για περισσότερο συντονισμό ε, εφαρμογής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ελπίζουμε ότι τότε δεν θα μας κατηγορήσουν ότι οι Βρυξέλλες έχουν πάρα πολλές εξουσίες, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει έναν ηγετικό ρόλο. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό στο πλαίσιο της πολιτικής και οικονομικής συγκυρίας, δεδομένου ότι όπως γνωρίζετε υπάρχει μεγάλη πίεση στους οικονομικούς πόρους για να το πω ευγενικά. Ε, για τις ε, προκλήσεις που έχουμε ε, για το διαδικτυακό εμπόριο θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε την επιβολή, την εφαρμογή της νομοθεσίας με ψηφιακά μέσα που θα δίνουν τη δυνατότητα καλύτερης ανταπόκρισης και καλύτερη συμμετοχή των εμπόρων και των καταναλωτών. Πρέπει μάλιστα οι σχετικές νομοθεσίες να συντονιστούν σε μεγαλύτερο βαθμό και περιμένουμε αναθεώρηση του κανονισμού CPC ε, που μέχρι το τέλος του 2014 για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς συντονισμού μας. Επίσης θα υπάρξει δημόσια διαβούλευση πριν από το καλοκαίρι για το θέμα αυτό. Ως το θέμα τώρα της ε, αποζημίωσης, ε, ε, οι μηχανισμοί εναλλακτική επίλυσης και διαδικτυακής επίλυσης των μηχανισμών είναι ένα, πάρα πολύ, ορόσημο για τη βελτίωση των ψηφιακής αγοράς. Γνωρίζετε ότι στις 12 Μαρτίου επιβεβαιώσαμε σε πρώτη πρώτη ανάγνωση και πριν από δύο μέρες το Συμβούλιο ενέκρινε, το ενέκρινε ε, και εκείνο, είναι ένα μεγάλο βήμα για τους καταναλωτές ε, σε όλη την Ένωση που θα μπορούν να επιλύουν έξω ε, δικαστικά τις διαφορές τους γρήγορα και αποτελεσματικά. Και επίσης οι έμποροι δεν θα έχουν το κόστος της επίλυσης των διαφορών, κάτι το οποίο ελπίζουμε να ενθαρρύνει την εμπιστοσύνη και των καταναλωτών και των εμπόρων στην ψηφιακή αγορά. Ε, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους, ε, τους, ε, τον Λούι Γκρέκ, ο οποίος είναι τώρα Υπουργός Υπουργαϊκών Υποθέσεων στην ε, Μάλτα και να σας ευχαριστήσω και εσάς ε, κύριε Πρόεδρε για την ε, δέσμευσή σας και την αποσύνση σας γιατί πραγματικά ήταν άνευ προηγουμένου μια τόσο γρήγορη και ισορροπημένη συμφωνία. Δεν έχουμε τελειώσει βέβαια. Θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο φιλική προς το χρήστη να είναι αυτή η εναλλακτική επίλυση και διαδικτυακή επίλυση μηχανισμών. Θέλουμε να υπάρξουν κατευθυντήριες γραμμές, θα τις υποβάλουμε και επίσης θα προβούμε και σε κάποια μέτρα για την ε, προώθηση αυτών των μηχανισμών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, όσον αφορά τώρα τις ε, συλλογικές αποζημιώσεις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε πάρα πολύ επικοδομητική επιρροή στις συζητήσεις. Γνωρίζω τις διάφορες απόψεις των οργανώσεων των καταναλωτών των εμπλεκομένων φορέων και των κρατών μελών. Αποτελεί η ισχυρή πεποίθησή μου ότι χρειάζεται ένα συνεκτικό πλαίσιο για το θέμα αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει πρωτοβουλία σε σχέση με το θέμα αυτό κατά το τρέχον έτος και ε, Ελπίζω να υπάρξει συνεργασία με τους συναδέλφους Αλμούνια και Ταγιάννη. Μπορεί η πρωτοβουλία αυτή να μην ε, ικανοποιήσει τις προσδοκίες όλων, αλλά είναι, ένας πάρα πολύ, είναι ένα πολύ καλό βήμα ε, σε ένα πάρα πολύ δύσκολο και ευαίσθητο θέμα. Ε, τώρα, η ενσωμάτωση των, των δικαιωμάτων των καταναλωτών ε, ε, στην ε, ψηφιακή ατζέντα. Και στις τομεακές πολιτικές υπάρχει το θέμα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ενέργεια, μεταφορές, τρόφιμα, ε, αηφόρος, ε, κατανάλωση. Εγώ συνεργάζομαι με τους ε, συναδέλφου μου για να εξασφαλίσω το γεγονός ότι αυτά τα στοιχεία λαμβάνονται υπόψη. Για παράδειγμα, με τον Επίτροπο Μπαρνιέ ολοκληρώνουμε μια νομοθετική πρωτοβουλία για του τραπεζικού λογαριασμού που θα προσπαθήσουν να βελτιώσει τη διαφάνεια και συγκρισιμότητα των τελών ε, για τους τραπεζικούς λογαριασμούς, ε, μείωση των εμποδίων, ε, όπως επίσης και άρση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες στην πρόσβαση στις τραπεζικές υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Ελπίζω λοιπόν ότι θα ολοκληρωθεί αυτό σύντομα. Όσον αφορά τώρα την οδηγία για τις πιστώσεις των καταναλωτών, θα δημοσιεύσουμε μία έκθεση για την εφαρμογή την καταναλωτική πίστη. Ε, η έκθεση θα γίνει από εξωτερικούς ε, αναδόχους. Θα υπάρξει μάλιστα και ε, πλήρης ενημέρωση στην Ιρλανδία, στην Ισπανία, στην Κύπρο για το θέμα της καταναλωτικής πίστης. Για τις συντάξεις οργανώνουμε, προετοιμάζουμε ένα έγγραφο που θα χρησιμοποιηθεί ως βάση διαβούλευσης με στόχο να αναγνωρίσουμε πώς θα μπορούσε μια συντονισμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση να βελτιώσει το, τη θέση των καταναλωτών ε, σε σχέση με τα συνταξιδοτικά ταμεία. Είδαμε επίση τα αίτια και τι συνέπειε ε, ε, υπερβολ... του υπερβολικού χρέους, γιατί έχουν γίνει πολύ εύκολα τα δάνεια για να δούμε πώς είναι η κατάσταση σε κάθε κράτο μέλος και να εντοπίσουμε τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε για να ανακοφίσουμε τον αντίκτυπό της. Περιμένουμε τα πορίσματα τη μελέτης που θα μα βοηθήσει να δούμε τι ε, δράση πρέπει να αναλάβουμε. Γίνεται επίσης διάλογος ε, πολυμερής που επικεντρώνεται στην ηλεκτρονική τιμολόγηση και πώς μπορεί κανείς ε, να βελτιώσει την ενεργειακή διαχείριση των καταναλωτών. Και τέλος, στο θέμα της ψηφιακής τεχνολογίας, ε, θα δημοσιεύσουμε τα πορίσματα μιας νέας μελέτης για την πρόσβαση και παροχή υπηρεσιών στο διαδίκτυο από την πλευρά, την οπτική γωνία των καταναλωτών. Και αυτό ε, θα μας δείξει τι χρειάζεται ακόμη να, κάνει, να κάνουμε για να ε, βελτιστοποιήσουμε ε, την πρόσβαση των καταναλωτών στις υπηρεσίες του διαδικτύου. Η δυνατότητά μας να εφαρμόσουμε σωστά την, την ατζέντα των καταναλωτών θα περάσει από το πρόγραμμα ε, για τους καταναλωτές και από τις διαπραγματεύσεις ε, για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο ε, εμείς έχουμε πάντοτε ως βασικό μας μέλημα την προστασία των καταναλωτών στο πλαίσιο μιας ψηφιακής ατζέντας. Ευχαριστώ πολύ. Well, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πληρέστατη η επισκόπηση αυτή. Σημείωσα πολλά για δραστηριότητες που ζητούσαμε εμείς ε, να υιοθετήσετε. Βέβαια για μας θα είναι πρόκληση να απαντήσουμε σε όλα αυτά, αλλά με χαρά να το κάνουμε. Οχτώ έχουν εγγραφεί, εννέα, ε, συνάδελφοι δέκα, άλλος κανείς. Μισή ώρα έχουμε θυμίζω, έτσι. Λοιπόν, νομίζω να ενισχύσουμε με την κυρία Γκέπχαρτ και τον κύριο Σφαμ. και δεν ξέρω από τις άλλες πολιτικές ομάδες η κυρία Ρούλε με τη σειρά. Η κυρία Γκέπχαρτ, ο κύριος Σφαμ. Για αλλαγή θα δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Γκέπχαρτ γιατί ήταν και η συγκήτριά μας για τον τραπεζικό λογαριασμό και θέλει πάρα πολύ... Τη... Βλέπω ένα πλατή χαμόγελο έχει φωτίσει το πρόσωπό της. Μετά ο κύριος Φαπ και οι υπόλοιποι. Παρακαλώ σύντομα να μιλήσετε. Αλλιώ θα έρθει ο κύριος Σταγιάννη και δεν θα προκάνουμε. Η Εύελεν. Ευχαριστώ. Ε, Μάλκομ. Καλώς ορίσατε κύριε Βόρτ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν όντως εκτενέστατη η παρουσίασή σας και πολύ ε, κατανοητή και πολλά υποσχόμενη. Εγώ τώρα θα ήθελα να απαντήσω σε πάρα πολλά θέματα, αλλά για αλλαγή δεν θα πω τίποτα για τις συλλογικέ αποζημιώσεις και αγωγές, γιατί ξέρω ότι θα τον φέρει ο Μάρκ Ταραβελά, αλλά ε, ε, να αναφερθώ σε άλλα θέματα. Αυτό που είπε ο Μάλκομ τώρα, ε, η πρόσβαση σε ένα τραπεζικό λογαριασμό. Αυτή είναι μια πρωτοβουλία και δική μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, με μια έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας γιατί είναι ένα πρόβλημα πάρα πολύ πιεστικό και δεσμεύτηκε και ο κύριος Μπαρνιέ τότε ότι γρήγορα θα φέρει ένα τέτοιο μέτρο. Ναι, πώς το περιμένουμε ακόμα παρακαλώ, μπορείτε να μου πείτε. Κανονικά περιμέναμε από το Φλεβάρι, το αργότερο το Μάρτιο να φέρετε την πρόταση έχετε κανένα νέο, πότε υπολογίζετε ότι θα τη φέρετε. Οι πολίτες πραγματικά το περιμένουν, τους ενδιαφέρει. Ένα δεύτερο, αναφέρατε μια εκστρατεία, μια καμπάνια για τα δικαιώματα των καταναλωτών. Και σε διάφορα κράτη-μέλη θέλετε να τη διοργανώσετε και μου φαίνεται και πολύ ωραίο. Μήπως θα είχε όμως νόημα, κύριε Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια στιγμή να κοιτάξει τα δικαιώματα που κατοχυρώσαμε για τους καταναλωτές και τους πολίτες ε, τα τελευταία χρόνια. Μπορούμε να εντοπίσουμε, όπως το κάναμε τον κύριο Μπαρνιέ για τα δέκα σημαντικότερα ερωτήματα, μπορείτε να κάνετε κάτι αντίστοιχο για τα δικαιώματα των καταναλωτών, για τους Ευρωπαίους πολίτες, άνδρες και γυναίκες, γιατί αυτό θα είχε πάρα πολύ νόημα, για να μπορέσουμε να προβάλλουμε αυτή την Ευρώπη μας και να την κάνουμε πιο κατανοητή για τους πολίτες. Γιατί πολύ συχνά Τα περισσότερα είναι που πρέπει πρώτα να μεταφερθούν στα κράτη-μέλη και μετά ο κόσμος τα αντιλαμβάνεται ως εθνικό δίκαιο. Μα όλα αυτά που κάνουν τη διαφάνεια είναι ευρωπαϊκό δίκαιο και προς όφελος των πολιτών και των καταναλωτών όσο και καταναλωτριών. Αυτό μπορούμε να το προβάλλουμε, να το διαφημίσουμε στα μάτια των πολιτών ο κύριος Σφάπ και μετά ο κύριος Μπουσόη και θα απαντήσει ο Επίτροπος στους τρεις πρώτους. Ο κύριος Σφάπ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, και εγώ χάρηκα πάρα πολύ για ε, τη δέσμευσή σας και την προσήλωση που δείχνετε στον πρώτο κιόλας μήνα ε, από την ανάληψη των καθηκόντων σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που ενδιαφέρεστε για την υλοποίηση, για την επιβολή και εφαρμογή των ήδη ηλυμένων αποφάσεων, γιατί φαίνεται και χωλαίνει σε πολλές περιπτώσεις η κατάσταση. Η οδηγία για τα ιατρικά προϊόντα, παράδειγμα, και εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βελτίωσε, τουλάχιστον η πρότασή της, ε, τα πράγματα. Το ίδιο ισχύει και για την εποπτεία των αγορών. Πολύ ε, καλά τα καταφέρετε με τη Γενική Διεύθυνση Βιομηχανία να κάνετε μια συμβαστική πρόταση και ασφάλεια των προϊόντων, ε, όλα αυτά ρυθμίζονται ωραία. Θα επανέλθω σε αυτό που μόλις ανέφερε η συνάδελφος η κυρία Γκέπχαρτ. Είναι θετική πρόταση. Πραγματικά πρέπει να το συζητήσουμε περισσότερο και να προβάλλουμε τι επιτύχαμε. Και λιγότερο ή τουλάχιστον εξίσου να συζητάμε ε, τι απομένει ακόμα. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε για να προωθήσουμε αυτή την υπόθεση της υλοποίησης και επιβολής του νόμου ε, στα κράτη-μέλη. Γιατί ε, στο θέμα τώρα των, ε, της καταλληλότητας των δρόμων, των αυτοκινητοδρόμων και των οδοστρωμάτων, τα κράτη-μέλη επειδή έχουν οδηγία για να είναι στο χέρι τους πώς θα το ρυθμίσουν. Μήπως εσείς θέλετε να κινηθείτε προς ένα κανονισμό για να είναι πιο ενιαία τα πράγματα αυτά και να μπορούμε να τα ελέγχουμε καλύτερα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπουσόη και μετά τα Ραμπέλα, Χάνσλικ και Ροσφόρ, για την Ροσφόρ, η επόμενη. Yes, I will be very brief, even the time very... Θα είμαι πολύ σύντομος, γιατί θέλω να ξεκινήσουμε και με τον κύριο Ταγιάννη ακριβώς στις 4. Είμαι εισηγητής εκ μέρους της Επιτροπής μας για την οδηγία περί Έχω ήδη συντάξει γνωμοδοτησία για την Επιτροπή ΕΜΚΟ και ξέρω ότι πρόσφατα εγκρίθηκε, όπως θα ξέρετε εγκρίθηκε προσφατοποιημένη πρόταση ε, της οδηγίας περί διαφάνειας, λαμβάνοντας υπόψη πολλές από τις τροπολογίες και το Κοινοβουλίου και της δικής μας της Επιτροπής. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία για το Κοινοβούλιο έχει φτάσει σε μπλοκάρισμα στο Συμβούλιο. Επίτροπε, έχετε καμία ε, είδηση από το Συμβούλιο για την ε, επόμενη φάση σε σχέση με την πρόταση αυτή και τι μέτρα θα λάβετε για να διευκολύνετε την επίτευξη συμφωνία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων για αυτή την οδηγία. Έπειτα, επόμενη ερώτηση για ένα θέμα που έχει να κάνει με την ε, παράλληλη εξέταση του θέματος της προστασίας των καταναλωτών και της υγείας, δηλαδή τις ιατρικές συσκευές. Έχει προταθεί ένας κανονισμός προκειμένου να ορίζονται όλοι οι όροι που θα πρέπει να αφορούν τις ιατρικές συσκευές μέχρι να τεθούν στην αγορά. Θα πρέπει τις ίδιες διαδικασίες να τις προβλέψουμε όπως και για τα φάρμακα Μιλάμε για τελείω διαφορετικά προϊόντα βέβαια. Δεν είναι τα ίδια τα διπλώματα ευρεσιτεχνία. Σε μερικέ περιπτώσει δεν υπάρχουν καθόλου και οι ιατρικέ συσκευέ έχουν πολύ διαφορετικό αντίκτυπο στου καταναλωτέ, του ασθενεί από τα φάρμακα. Είναι πολύ διαφορετικέ οι δυναμικέ τάσει τη αγορά. Ποιε είναι οι προθέσει σα λοιπόν για να έχετε καλύτερη συνεννόηση με το Κοινοβούλιο και ποια είναι οι διαφο... ως προς τις διαφορές των δύο κατηγοριών προϊόντων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Γκέμπχαρτ είπε ότι υποσχέθηκα πολλά. Δεν νομίζω ότι υποσχέθηκα πράγματα που δεν μπορούμε να πετύχουμε. Διότι τα τελευταία 30 χρόνια είμαι στον πολιτικό βίο και ξέρω τι θα πει δίνω υπόσχεση. Σημαίνει ότι κανείς πρέπει να κρατάει και αυτά που έχει πει. Έχω υποσχεθεί λοιπόν πολλά, γιατί είμαι βέβαιο ότι πολλά θα πετύχω, όπω την οδηγία για, την, για τα τραπεζικά που τελικά εξετάστηκε 6 εβδομάδε νωρίτερα. Όταν μίλησα λοιπόν για τι τραπεζικέ υπηρεσίε και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα, είπα ότι δεν ήταν το δικό μου σφάλμα ούτε του κυρίου Μπαρνιέ που υπήρξε καθυστέρηση στην αρχή τη διαδικασία. Ήδη όμω προβλέπονται συζητήσει τον ερχόμενο μήνα και θα γίνει και ανακοινωθέν στο, στον τύπο για την έναρξη εξέταση τη οδηγία. Θα είναι λοιπόν πρωτοφανέ, εάν δεν γίνει αυτό τον ερχόμενο μήνα. Κατά 99% θα έλεγα το Μάιο θα αρχίσει η εξέταση. Φαντάζομαι ότι θα εγκριθεί μετά από το σώμα των Επιτρόπων και νομίζω ότι αυτό ήταν που θέλατε κι εσείς αφού εργαστήκατε τόσο σκληρά. Για μια χάρτα των δικαιωμάτων των καταναλωτών και εγώ είμαι υπέρ της ιδέας αυτής, ιδίω τώρα που έχουμε συνηθίσει στην ενιαία αγορά βέβαια. Είναι εκπληκτικό πως πολλές φορές προέρχονται ακόμα επιχειρήματα από εκεί που δεν το περιμένουμε για την ε, άρση των φραγμών, ε, την ελπίδα τους αντιμετώπιση κάθε φορά που γίνεται μια πρόταση. Τώρα βέβαια βλέπουμε ότι κάθε φορά που κάποιος παραβιάζει τον νόμο σε μια χώρα, αυτό επηρεάζει ολόκληρη τη χώρα. Βεβαίω, αυτό για την ενιαία αγορά δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να πάψουμε να επιδιώκουμε να τη δημιουργήσουμε. Όχι, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τι παραβιάσει του νόμου και να είμαστε βέβαιοι ότι το δίκαιο ισχύει παντού. Το ίδιο με το Σέγγεν. Για τι χώρε που έχουν αποδεχτεί να συμμετάσχουν, δεν σημαίνει ότι θα το καταργήσουμε γιατί κάποιο με ποινικό μητρό μετακινείται από μια χώρα στην άλλη. Όχι, οι έλεγχοι πρέπει να ενταθούν. Πρέπει να υπάρξει καλύτερη επιβολή των νόμων και καλύτερη επικοινωνία. Νομίζω και η ενιαία αγορά είναι ακρογωνιαίος λίθος τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ακριβώ το ίδιο ισχύει όπω και για το χώρο Σέγγεν. Εδώ ένα σχόλιο και για το πώ μπορούμε να ενδυναμώσουμε την ενιαία αγορά. Εργαζόμενοι προ αυτή την κατεύθυνση και δημοσιοποιώντα, προβάλλοντα ε, τα ωφέλη για του καταναλωτέ και ω προ τι ανταγωνιστικές τιμέ και ω προ τη διαθεσιμότητα προϊόντων, ιδίω στι χώρε που γνωρίζω καλύτερα, από τη στιγμή που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε άμεσος αντίκτυπος ως προς τη σύγκριση των τιμών και χάρη στο ενιαίο νόμισμα αλλά κυρίως χάρη στην ενιαία αγορά. Αλλά υπήρξε και αύξηση του ζωτικού επίπεδου. Και κυρίως μπορεί κανείς να ψωνίζει όπου θέλει και να έχει ευκολότερη πρόσβαση στα προϊόντα. Κύριος Μπουζόη, έκανε ένα εύστοχο σχόλιο για τις ιατρικές συσκευές. Στο πρώτο μέρος τη ερώτηση θα είχα να πω το εξή. Κάποτε ήμουν υπέρ του κυρίου, τάχθηκα υπέρ του κυρίου Ταγιάννη στο Συμβούλιο και αυτό συζητήθηκε. Έκτοτε, με τον κύριο Ταγιάννη δεν το ξανασυζητήσαμε, αλλά ξέρω ότι θα έρθει στις 4 εδώ και εξ όσο γνωρίζω από εκείνη τη συνάντηση του Συμβουλίου του τουλάχιστον, ήταν ότι ήμουν ο μόνος που ακολούθησε αυτή τη στάση. Και για λόγους συναδελφικότητας, δεν ξέρω τι θα είχα κάνει αν έπρεπε να επιμείνω και να υπερασπιστώ την πρόταση αυτή. Διότι εξεπλάγει που ο καθένα ε, ήθελε αντέκρουε την πρόταση αυτή, λέγοντα ότι δεν θα έπρεπε να την καταψηφίσουμε. Η Επιτροπή θα έπρεπε να κάνει κάτι. Αυτό σα λέω ότι ήταν η αντίδραση που έλαβα βέβαια όταν ε, εκπροσώπησα τον κύριο Ταγιάννη και τον υπερασπίστηκα ενώπιον του Συμβουλίου. Βέβαια τώρα, αν κατάλαβα καλά το σχόλιο σα, Θέλετε μεταχείριση ανάλογη με τα φάρμακα. Συμφωνώ με αυτό. Ε, η πρόταση της Κομισιόν προς αυτή την κατεύθυνση κινείται. Η αγορά αυτή βρίσκεται σε άνθηση και ως προς τις ανάγκες που έχουμε σε καιρός οικονομικής κρίσης είναι σημαντικό αυτό. Δίνει και ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε πολλές περιοχές του κόσμου. Οπότε ας μην κάνουμε τίποτα για να δυσκολέψουμε αυτό το μηχανικό κλάδο. Ε, ε, αφορά βέβαια αυτό το θέμα και την ασφάλεια των ασθενών, γιατί ασθενείς και κατανοητές εδώ συμπίπτουν. Είναι δύο κατηγορίες ανθρώπων που πρόκειται για την ίδια ομάδα ουσιαστικά εδώ. Ναι, θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος, ε, εξέταση πριν την είσοδο στην αγορά και μετά, αλλά η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι κατά του να απαιτείται για το υψηλό και συσκευέ πρώτερη έγκριση, πριν την είσοδο δηλαδή στην αγορά, με ε, δεσμευτικό χαρακτήρα. Ευχαριστούμε. Βλέπετε ότι ο χρόνο μα πιέζει. Ε, θα ζητήσω λοιπόν από του συναδέλφου να παραμείνουν σε ένα κέριο ερώτημα ο καθένα, γύρω στο ένα λεπτό, αν γίνεται. Νομίζω ότι μπορείτε να τα καταφέρετε. Ο κύριο Ταραμπέλα, η κυρία Χάνσλικ και ο κύριο Ρόσφορ. Θα σας χτυπήσω αν ε, καθυστερήσετε. Ευχαριστώ Πρόεδρε κύριε Επίτροπε. Η κυρία Γκέπχαρτ το μαρτύρησε αυτό που ήθελα να σας πω για τις ε, διαδικασίες συλλογικής αποζημίωσης και αγωγής. Σας ευχαριστώ που το αναφέρατε. Ε, κάθε επίτροπος που αναλαμβάνει αυτό το χαρτοφυλάκιο το βάζει στις προτεραιότητες του. 25 χρόνια το συζητάμε. Είχαμε πράσινες βίβλους και λευκές και ένα σωρό έγγραφα και ακροάσεις και έκτοτε μηδέν στο παρόλο που η διαδικασία αυτή σήμερα είναι επίκαιρη. Έχουμε ένα σωρό νέες αγορές, νέες τεχνολογίες, ε, κινητά τηλέφωνα, υπολογίστες, αυτοκίνητα, ε, αλλά και ιατροτεχνολογικά προϊόντα και σκευάσματα. Είδαμε διαρροές που υπήρξαν από εμφυτεύματα ε, στήθους. Ε, ξέρετε, λοιπόν υπάρχουν μια σειρά προβλημάτων και μπορούν από κοινού οι καταναλωτές να ενωθούν και να προχωρήσουν σε συλλογική δράση και αγωγή για αποζημίωση. Το είπε και η κυρία Ρέντινγκ και ο κύριος Σαλμούνια συνεργάζονται, αλλά η κυρία Ρέντινγκ όταν τη ρωτήσαμε, τις 5 Μαρτίου συγκεκριμένα, σε κοινοβουλευτική ερώτηση. Τελειώνω, Πρόεδρε. Μία πρόταση έχω πει. Εσέβομαι το ένα λεπτό. Είπε η κυρία Ρέντιγκ ότι το σκέφτεται. 25 χρόνια μας προβληματίζει αυτό. Ε, δεν θα καταλήξουμε ποτέ. Εντάξει, πιστεύουμε, μας δίνει το λόγο σας, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να έρθει αυτή η πρόταση και πιο ε, Πότε έχει προχωρήσει έχει δρομολογηθεί στο pipeline που το λέτε εκεί στην Κομισιόν. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάντσλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη, αλλά θα ξεπεράσω το λεπτό, γιατί έχω τρεις πολύ σημαντικές ερωτήσεις να κάνω. Για την οδηγία για τα προϊόντα καπνού που συζητούμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, το ηλεκτρονικό τσιγάρο περιέχει νοικοτήνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε κάποια οριακή τιμή. Και όταν ξεπερνούν αυτό το όριο, ε, τα τσιγάρα αυτά θα θεωρούνται ιατρικά προϊόντα και βάσματα σαν φάρμακα. Και ε, γίνονται και προτάσεις μέχρι να απαγορευθούν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, τέτοια απειλή απαγόρευσης. Και πώς μπορεί μια εταιρεία να λάβει άδεια βάσει τις οδηγίες. Ε, ερώτηση δεύτερη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αποτρέπει τους νέους από το να αρχίζουν το κάπνισμα. Ε, τι ε, φρονείται για τα νεωτερικά προϊόντα καπνού, νοτόμα. Τρίτη ερώτηση. Τι γίνεται με τις καπνοβιομηχανίες και τις καλλιέργειες. Ορισμένες χώρες θα πληγούν περισσότερο από τις αλλαγές. Θα τα λάβει όλα αυτά υπόψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Ζωσφό. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που στο τέλος μιλήσατε για τον προϋπολογισμό. Μάλιστα εδώ θα έχετε την υποστήριξη για τον προϋπολογισμό αυτό για την προστασία των καταναλωτών που είναι από τους χαμηλότερους προϋπολογισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη όμως σε αντάλλαγμα περιμένουμε να μας υποστηρίξετε για να μπορέσουμε να καταλήξουμε με το Συμβούλιο σε αυτό το καθόλου θέμα. Θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή σε ένα θέμα που σπανίως αναφέρεται με Αι. Είναι τέτοια οικονομική κρίση στην Ένωση που αλλάζουν ε, οι ε, καταναλωτικές συνήθειες των Ευρωπαίων με νέες συνήθειες, με ανταλλαγή προϊόντων. Ε, το c του από καταναλωτή σε καταναλωτή, μεταχειρισμένα προϊόντα, ρούχα, ε, πληστηριασμοί στο διαδίκτυο και αλλού. Αλλάζουν λοιπόν οι καταναλωτικές συνήθειες, ε, αναδύονται καινούριε και δεν θα πρέπει να μειώνεται, να υποβαθμίζεται η προστασία του καταναλωτή. Ε, όλες οι προτάσεις μας ε, αφορούν την κλασική προστασία του κλασικού καταναλωτή που αγοράζει ένα προϊόν κτλ. Έχουμε όμως νέα φαινόμενα τώρα στους καιρούς της κρίσης. Τα λαμβάνετε αυτά υπόψη σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα παρακαλέσω τώρα τον Επίτροπο να απαντήσει, αλλά πριν το πράξω πρέπει να σας πω να ετοιμάζετε με σύντομες ερωτήσεις η επόμενη. Κοράτσα, Μπίλτ, Στάιλερ και Άριας. Παρακαλώ. Για τι συλλογικέ αγωγές και αποζημιώσεις μπορώ να σας πω το εξή. Ε, οι υποσχέσει μου είναι μόνο αυτές που μπορεί να γίνουν πραγματικότητα. Το να μην κάνουμε τίποτε δεν αποτελεί επιλογή. Εγώ είμαι εδώ πέντε μήνες και δεν μπορώ να πω τι, τίποτα για τα 25 χρόνια, αλλά μπορώ να σας πω, επειδή έχω τι σωστές πληροφορίε στη διάθεσή μου, ότι θα υπάρξει μια πρωτοβουλία φέτος, Τώρα ποια ακριβώς μορφή θα λάβει αυτή η πρωτοβουλία, αυτό ακόμη το συζητούμε ε, στο Σώμα των Επιτρόπων. Ελπίζουμε όμως να υπάρξουν εξελίξεις κατά τις ερχόμενες εβδομάδες για να πούμε ακριβώς τι πρωτοβουλία θα είναι αυτή. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι ό,τι και να κάνουμε θα έπρεπε οπωσδήποτε να οδηγηθούμε σε νομοθεσία για το θέμα αυτό. Εγώ κατά την ε, ακρόασή μου είχα πει ότι είμαι υπέρ ε, της ε, συλλογικής αποζημίωσης. Ε, ψήφισα υπέρ και όλα στο δικό μας κοινοβούλιο όταν είχαμε συζητήσει αυτό το θέμα, περάσει νομοθεσία για το θέμα αυτό. Βέβαια μερικές φορές στην πολιτική πρέπει να είμαστε υπομονετικοί και να κάνουμε μικρά βήματα προς ένα στόχο, αρκεί όμως τα βήματα αυτά να είναι προς τα μπρος και προς τα πίσω. δεν θα υπάρξει μια τροπολογία δεν ε, θα, θα είναι κάτι ουσιαστικό, κάτι αισιόδοξο, ε, δεν θα είναι απλώς νεκρές ιδέες. Βέβαια, Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές όταν περιμένει κάτι, κάτι πολύ καιρό, μετά δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του. Όσον αφορά τώρα τα προϊόντα καπνού και τις οικονομικές συνέπειες, το ηλεκτρονικό τσιγάρο υπάρχει ήδη στην αγορά. Το καλύτερο είναι να ε, υπάρξει ρύθμιση όσο το δυνατόν καλύτερη, παρά το γεγονός ότι συμφωνώ μαζί σας, τουλάχιστον αυτό κατάλαβα ότι είπατε, ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο μπορεί να δώσει μια λανθασμένη εντύπωση ασφάλειας στους καπνιστές ή πρώην καπνιστές, γιατί πιστεύουν ότι δεν καπνίζουν πια, γιατί καπνίζουν ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο και ότι δεν υπάρχει καπνό εκεί. Αλλά βέβαια οι συνέπειες είναι επίσης επιβλαβείς ε, για την υγεία τους ε, και αν ήθελα να αρχίσω μία εκστρατεία, θα αρχίσω μία εκστρατεία για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα συγκεκριμένα. Θα ήθελα λοιπόν να ε, υπάρχει ένα κατώτατο όριο, αλλά δεν θα ήθελα να υπάρξει υπερβολική ρύθμιση. Η τρέχουσα οδηγία για τον καπνό έλαβε ιδιαίτερη υποστήριξη σε τέτοιο βαθμό ώστε ο εισηγητής της ΕΜΒΗ προτείνει περαιτέρω ε, περιορισμούς όπως ε, απλά ε, γενικής φύσεως τυποποιημένα πακέτα κλπ. Βέβαια από την άλλη πλευρά στο Συμβούλιο δεν θα είναι πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα. Ε, εντάξει δεν θα είναι εύκολα ούτε εδώ αλλά δεν θα είναι εύκολα ούτε στο Συμβούλιο. Ειδικό κυρίως γιατί υπάρχουν κάποια εθνικά ζητήματα όπως τα τσιγάρα, τα λεπτά, τα slim, ε, τις ε, ουσίες, ε, τις, τις αρωματικές, τις ορισμένα τέλος πάντων κάποια προϊόντα καπνού που έχουν κάποιο περιφερειακό χαρακτήρα, για να το πω έτσι. Το βασικό ζήτημα όμως για τους υπουργού Οικονομικών είναι το θέμα των ε, χρημάτων και των ε, θέσεων απασχόλησης. Κοιτάξτε, ε, δεν θέλω να γίνω κακός, αλλά προσπαθούμε να μειώσουμε τον αριθμό των καπνιστών. Όταν έχουμε λοιπόν ένα στόχο τέτοιο, πρέπει, να μειώ... πρέπει όντως αυτό να θέλουμε να, ε, να το έχουμε ως στόχο. Θέλουμε να το μειώσουμε 2% ας πούμε σε μια περίοδο πενταετή, δηλαδή περίπου 2,4 εκατομμύρια καπνιστές λιγότερα, λιγότερους το χρόνο. Τώρα κατά πόσο αυτό θα έχει επιβλαβείς συνέπειες οικονομικές για κάποιες χώρες, ναι θα έχει. Αλλά θα έχει και θετικές οικονομικές συνέπειες, γιατί τα χρήματα που θα εξοικονομήσουμε από τους πρώην καπνιστές θα επενδυθούν σε άλλα, ε, σε άλλους τομείς της οικονομίας, δημιουργώντας ενδεχομένως περισσότερες θέσεις απασχόλησης από αυτές που χάθηκαν. Κοιτάξτε, και πάλι δεν θέλω να γίνω δυσάρεστος, αλλά αν έπαιρνα το επιχείρημά σας, το επιχείρημα που παραθέσατε, που είναι που είπατε ότι είναι και τις καπνοβιομηχανίες, δεν λέω ότι είναι αυτή η άποψή σας, αλλά πάση περιπτώσει λέτε τι λένε οι άλλοι. Τότε ότι, ότι θέλω να να ότι κανείς μπορεί να προωθήσει τον καπνό και με αυτή την έννοια η οικονομία θα ενθαρρυνθεί επίση. Ναι, πρέπει από τη μία να καταπολεμήσουμε το κάπνισμα, γιατί ξέρουμε ότι το κόστος για τις κυβερνήσεις είναι δισεκατομμύρια. Αν θέλουμε να επιτύχουμε το στόχο μας, θα, θα εξοικονομήσουμε ε, πάρα πολλά χρήματα σε νοσοκομεία, γιατρούς, ε, ε, οπότε... Θα υπάρξει πλήγμα. Ναι, βεβαίως θα υπάρξει πλήγμα, αλλά νομίζω ότι ε, και το όφελος θα είναι σίγουρα μεγαλύτερο ίσο του πλήγματος. Οπότε η ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή, ναι, βεβαίω θέλει να επιτύχει του στόχου μείωση του καπνίσματο και να υπάρξει μια σωστή, να τη σωστή ισορροπία τέλο πάντων στα διάφορα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τώρα τι τάσει κατανάλωση που τι ανέφερε ο κύριο Ροσφόρ στο πλαίσιο του προγράμματος για τους καταναλωτές, Μία, ένα ερώτημα με είχε απασχολήσει εμένα σε μία διάσκεψη ΜΚΟ. Ναι, λειτουργία ψηφιακής αγοράς, προστασία καταναλωτών. Σε μερικέ χώρε όμως δεν υπάρχει τίποτα να καταναλωθεί. Ναι. Οπότε το ερώτημά μου είναι, Χρειαζόμαστε περισσότερη νομοθεσία, περισσότερη προώθηση, ναι, περισσότερη προώθηση καταναλωτικών δικαιωμάτων σε περίοδο κρίση. Γιατί γίνεται πιο ευάλωτο ο καταναλωτή όταν αρχίζει η κρίση. Ποιο θα υποφέρει περισσότερο από την κρίση, από την οικονομική κρίση ε, στον καταναλωτικό κόσμο. Θα είναι οι πιο ευάλωτοι λόγω ηλικία, λόγω κατάσταση ε, ε, και βεβαίω επειδή θα υπάρξουν απάτε, επειδή θα υπάρξουν νέε τέλο πάντων οι οποίες θα μπορούσαν να επιδεινώσουν το ευάλωτο των καταναλωτών. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να επαγρυπνούμε ακόμη περισσότερο για τα δικαιώματα των καταναλωτών σε περίοδο κρίσης. Γιατί η κρίση προσθέτει στο ευάλωτο των καταναλωτών. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενες τρεις σύντομες ελπίζω ερωτήσεις, Κοράτσα Μπίλ, Τεστάιλερ και Αρίας. Κυρία Κοράτσα Μπίλτε, επειδή πρέπει να φύγετε. Ευχαριστώ. Υπάρχει πρόβλημα με την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ε, τροφική αλυσίδα. Βλέπουμε έναν εθνικό υπερβολικό προστατευτισμό ε, για την παραγωγή τροφίμων και αυτό ανησυχεί τον κόσμο, ιδίω μετά το σκάνδαλο με το αλλαγήσιο κρέα. Τι θα κάνει αποτελεσματικά και γοργά η Επιτροπή με το πρόγραμμα δράση για να αντιμετωπίσει το σκάνδαλο του ο κρέατο. Έχω τρία ερωτήματα λοιπόν. Πρώτα απ' όλα, εχνηλησιμότητα. Στο πρόγραμμα δράση μιλάτε για επιτάχυνση τη έγκριση, τη έκθεση για την υποχρεωτική ετικετοθεσία για το κρέα, για οποιοδήποτε προϊόν κρέατο. Και ήμουν εγώ υπεύθυνη ηγέτρια για το θέμα αυτό και την ανάλογη ετικετοθεσία. Με ενδιαφέρει λοιπόν ιδιαίτερω να ακούσω τι απόψει σα. Έχετε απάντηση για την απέτηση αυτή των καταναλωτών για μεγαλύτερη λασιμότητα. Έπειτα, υπάρχει νομοθεσία που να είναι ανώδυνοι και να μπορούν να πούν οι εταιρείε ότι δεν το ξέραμε, μα συγχωρείτε γιατί δεν ξέραμε τι κάνουν οι προμηθευτέ μα. Ποιο είναι υπεύθυνο, ποιο είναι υπέτειο ενώπιον των καταναλωτών. Στην αναθεώρηση που προγραμματίζεται για το ποινικό δίκαιο και το... για τι ποινικέ κυρώσει και του ελέγχου με την οδηγία 82-2004 θα ενισχυθούν εδώ τα πρόστιμα, θα υπάρξουν κυρώσεις, θα υπάρχουν περισσότεροι έλεγχοι και δοκιμές. Αρκεί αυτό κάτι που θα αφορά μόνο τους μικρούς παραγωγούς που θέλουν να έχουν πρόσβαση στις αγορές, πώς θα διευκολυνθούν αυτοί. Η πρόθεση παραβίασης της νομοθεσίας της, για την τροφική αλυσίδα ε, είναι κάτι που μπορεί να εντοπιστεί, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, μπορεί να είναι αρκετό κριτήριο. Κάτι τελευταίο, Πρόεδρε, ευχαριστώ για την απάντηση που δώσατε στο κρατό μου ερώτημα για το θέμα της Ήθελα να σα καλέσω, καλέσω και πάλι να το δείτε με τον βιομηχανικό κλάδο, διότι η αντίδραση πανικού ε, που, και διαστάσει που πήρε το θέμα με την απόσυρση των προϊόντων και, την, ε, και, το, το ότι πετάχτηκαν στα σκουπίδια πραγματικά ε, είναι σοβαρό γιατί είναι άλλο να λέμε ότι το πρόβλημα δεν ήταν θέμα επισήμανσης και άλλο να λέμε ότι δεν ήταν θέμα τροφική αλυσίδα. Εδώ λοιπόν κάτι έπρεπε να κάνετε με του κεφτέδε και τα λαζάνια και να πείτε σε όλου αυτού που πέταξαν τα τρόφιμα ότι τα πετάξανε τζάμπα. Έπρεπε να ενημερώσουμε του καταναλωτέ ότι δεν είναι θέμα ε, ασφάλεια των τροφίμων, είναι θέμα τικετοθεσία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει, είναι ως πρώτο αίτιο για τους πρώιμους θανάτους ε, την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών. Εδώ λοιπόν πρέπει να πω ότι σήμερα υποδέχτηκα καλεσμένο σε ένα σεμινάριο για την κατανάλωση νοπλωματοδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το τι μέτρα πρέπει να ληφθούν για την προστασία της δημόσιας υγείας. Με συμμετοχή από ιατρούς και ειδικού του χώρου. Είναι πολύ θλιβερό αυτό, παρόλο που η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων ε, Γεωργίας, Υγείας και Φορολογίας ήταν προσκαλεσμένη ε, στο, στην αίθουσα του σεμιναρίου, αλλά κανείς δεν προσήλθε. Αναρωτιέμαι λοιπόν, δεν θα έπρεπε κάποιο από τι υπηρεσίε σα να έχει έρθει η κυρία Τεστόριν εδώ ω επικεφαλή τη Γενική Διεύθυνση. Δεν θα έπρεπε να είναι κάποιο από το σεμινάριο. Είναι πολύ σημαντικό. Και το γεγονό ότι στη Σκωτία έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο εδώ με τις ε, ελάχιστες τιμές. καλό θα ήταν να ακούσετε και τη δική μας εμπειρία, διότι η σκοτσέζικη βιομηχανία στο χώρο αυτό έχει προσφύγει κατά της κυβέρνησης της ε, περιφέρειας αυτής. Μάλιστα, ε, μια επιπλέον πρόσκληση για σας. Ε, δεν θα προλαβαίνετε να έρχεστε. Ο κύριος Αρίας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ε, για τα όσα μας είπατε και για την εργασία σας. Ως ε, συντονιστής της ομάδας εργασίας για την ενιαία ψηφιακή αγορά θα ήθελα να σας πω ότι γίνεται πολύ καλή δουλειά για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Έχει κάνει αυτή τη στροφή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και ενημερώνει επιγραμμικά για τα δικαιώματα τους ε, πολίτες και τους καταναλωτές. Με ένα ιστότοπο για τα χαρακτηριστικά και τις τιμές ε, για τα προϊόντα. Πάρα πολύ καλή πραγματικά ε, αυτή η πρωτοβουλία που έχει ανάγκη το ψηφιακό περιβάλλον στην Ευρώπη. Αυτά δεν θα πρέπει μόνο να υπάρχουν αλλά και να λειτουργούν σωστά για να μην έχουν το αντίθετο ε, αποτέλεσμα. Η ε, επιγραμμική και εξοδικαστική επίλυση διαφορών είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική και για τους καταναλωτές και για τις μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις. Ερωτώ, ποιες άλλες πρωτοβουλίες λαμβάνετε εδώ, αναλαμβάνετε μάλλον, για να αυξηθεί η εμπιστοσύνη σε μια νέα ψηφιακή αγορά και τι θα κάνετε ε, για να είναι αποτελεσματικές αυτές οι δράσεις. Ευχαριστώ. Τελευταία ομάδα ερωτήσεων. Ελπίζω να προλάβουμε. Ε, Βάντερ Κάμπ. κάμπος. Ε, σας δίνω το λόγο για να απαντήσετε κύριε Επίτροπε πριν ακούσουμε τις τελευταίες τρεις ερωτήσεις. Θα ήθελα να αρχίσω με το θέμα του αλογίσιου κρέατος, γιατί αυτό είναι ένα ζήτημα καταναλωτικό, πράγματι. Είναι λοιπόν ε, η... το κατάλληλο φόρουμ να το συζητήσουμε. Ακόμη και όταν έγιναν όλα τα τεστ, όλοι οι έλεγχοι, οι έλεγχοι, τους έλεγχους πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Δεν μπορούσε όμως η Επιτροπή να υποχρεώσει τα κράτη-μέλη να, να κάνουν ε, τους ελέγχους αυτούς, παρά το γεγονός ότι κατά 75% το χρηματοδοτούμε ε, όλα τα κράτη-μέλη συνεργάστηκαν και περίπου το 1 τρίτο έκαναν και επιπλέον ελέγχους από αυτές που είχε συστήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και σας το λέω αυτό, η Γερμανία 256 τεστ ε, της ε, ζητήθηκαν και έκανε 358. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ελέγχθηκαν όλα τα σφαγιασμένα άλογα σε όλα τα σφαγεία. και άλλοι έκαναν ε, παρόμοια πράγματα και τα περισσότερα, πολλά κρατημέλη έκαναν και περισσότερα από αυτά που του ζητήθηκαν. Λοιπόν, αν θέλετε να με ρωτήσετε κατά πόσο έχουμε παρκή χνηλασιμότητα, ναι, θα έλεγα. Σας πω ένα παράδειγμα τα λαζάνια ε, με βοδινό που βρέθηκαν ε, στο ένα, σε ένα βρετανικό σούπερ μάρκετ ε, σε μερικές ώρες. Θα μπορούσε κανείς να πάει με τα ίχνη που άρχισε, που, ήταν, που, από πού ελήφθη το κρέας, πού έγινε η επεξεργασία του, πώς έγινε η διανομή και κατέληξε στο βρετανικό σούπερ μάρκετ. Το ερώτημα λοιπόν του κατά πόσο κάποιος θα έπρεπε να επεκτείνει την ετικετοθεσία ε, της προέλευσης ε, νοπού ε, βοδινού κρέατος, γιατί το ξέρετε ότι μετά θα πάει και στο εγωπρόβιο κρέας, θα επεκταθεί περαιτέρω κατά τους ερχόμενους μήνες. Το κατά πόσο θα έπρεπε λοιπόν να επεκταθεί και για το επεξεργασμένο κρέας, κοιτάξτε αυτό δεν είναι ένα ζήτημα ιχνηλασιμότητας, είναι καλύτερης διαφάνειας και καλύτερη, ζήτημα καλύτερης πληροφόρησης προς τον καταναλωτή. Όμως το ε, σκάνδαλο με το κρέας αλόγου θα είχε συμβεί ακόμη και αν είχαμε ε, το, την σήμανση της χώρας προέλευσης. Άρα ε, έχουμε λοιπόν, ε, επειδή υπήρχε τα τεστ του DNA, καταλάβαμε τι ακριβώς υπήρχε μέσα, αλλιώς θα ξέραμε ότι είναι άλογο. Δηλαδή ελέγχαμε για βακτήρια, αλλά δεν ξέραμε ε, πώς, γιατί ακριβώς κρέας μιλούσαμε. Ξέρουμε τώρα λόγω του DNA ότι ήταν τέλος πάντων ε, βοδινό κρέας, αλλά είχε μέσα και 20% άλογο. Ε, υπάρχουν αρκετοί ευρωβουλευτέ που είναι υπέρ αυτής της Το ευκολότερο είναι να πει κανεί ναι βεβαίω, θα προχωρήσω και θα το κάνω. Όμω πρέπει να περιμένουμε τη μελέτη αξιολόγηση αντικτύπου ο, ο στόχος ήταν το τέλο αυτού του έτου, είχε πει το Κοινοβούλιο. Ελπίζουμε η έκθεση να είναι έτοιμη μέχρι το τέλος του καλοκαιριού τρεις μήνες νωρίτερα δηλαδή και βάσει αυτής της έκθεσης ε, θα ε, δράσουμε. Υπάρχουν διαφορετικέ απόψει μεταξύ των κρατών μελών για το κατά πόσο θα έπρεπε να ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία. Υπάρχουν κράτη-μέλη που διαφωνούν γραπτώ, γιατί αυτό το θέμα είχε προκύψει και στο παρελθόν. Υπάρχουν κράτη-μέλη που είναι υπέρ. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη τα οποία ήταν κατά, αλλά τώρα είναι υπέρ. Αλλά αυτό συμβαίνει συχνά στην πολιτική. Πρέπει να δει κανείς και το διοικητικό φόρτο που σημαίνει κάτι τέτοιο. Όπως είπα και στην Επιτροπή, ε, στην Επιτροπή Πολιτισμού, έχω ένα... Ε, εγώ έχω... είμαι ανοιχτό ε, σε σχέση με το θέμα αυτό. Να δούμε ποιο θα είναι το διοικητικό άχθος. Είναι ευκολότερο να πει κανείς ότι αυτό το παιχνίδι, αυτό το πλυντήριο έγινε, κατασκευάστηκε στην Κίνα, στη Μάλτα ή στη Γερμανία και είναι δυσκολότερο να πει κανείς ότι ο κοιμάς ας πούμε γράφει στην ετικέτα ότι είναι λίγο ρουμανικός, λίγο μαλτέζικος, λίγο γερμανικός. Ε, θα πρέπει να γράφει που γεννήθηκε το ζώο, ε, που ε, έγινε η εκτροφή του, που σφαγιάστηκε κλπ. Τι προτείνουμε λοιπόν. προτείναμε ένα πακέτο το οποίο ακόμη δεν έχει εγκριθεί από το Σώμα των Επιτρόπων, αλλά ελπίζω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο τις ερχόμενες εβδομάδες, τέλος πάντων κατά πάσα πιθανότητα αυτό το μήνα ακόμη, θα συμπεριλάβει την υγεία των ζώων, των ε, φυτών, ε, όπως επίσης και το θέμα των ελέγχων. Θέλουμε να μην αρκούμεθα μόνο στο να λέμε, όπως λέμε στις οδηγίες, ότι οι ποινικέ κυρώσεις κάθε φορά που εγκρίνουμε μια νομοθεσία πρέπει να είναι αποτρεπτικές και κατάλληλες, αλλά πρέπει να πάμε πέρα από αυτό και να πούμε ότι και οι οικονομικές κυρώσεις πρέπει να αντικατοπτρίζουν το οικονομικό κέρδος, το κέρδος αυτών που έκαναν το έγκλημα. ε, το να λέει κάποιος ε, ότι είναι βόλιο κρέας κάτι ενώ είχε 20-30% κρέας αλόγου, αυτό το έκανε κανείς ε, γιατί υπάρχει οικονομικό κέρδος επειδή το ένα είναι πιο ακριβό απ' το άλλο, ε, τουλάχιστον τότε ε, η, πρέπει το έγκλημα, πρέπει η αξιόπινη πράξη, εν πάση περιπτώσει, να μην επιφέρει κέρδος. Έχει συμβεί και στο παρελθόν άνθρωποι που έκαναν ε, ε παραπλανητική ετικεφοσία ε, να συνεχίζουν να τιμωρούνται μεν προσωρινά αλλά να μην γίνεται καν αναστολή της αδειάς τους. Εν πάση περιπτώσει ε, αυτό πρέπει να σταματήσει. Η δεύτερη πρόταση που κάνουμε σε αυτό το πακέτο είναι να υποχρεώσουμε σε ελέγχους σε μερικές περιπτώσεις. Ε, στην περίπτωση του κρέας αλόγου πήγαμε πέρα από τους ε, ελέγχους που είχαμε προτείνει. Παραμένει βέβαια μία σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτές τις ειδικέ περιπτώσεις ε, που ανακύπτουν τέτοια ζητήματα, πρέπει να έχουμε την εξουσία να υποχρεώσουμε να γίνουν κάποιοι έλεγχοι. Στην περίπτωση τώρα της πατάλης των τροφίμων. Κοιτάξτε, εγώ ήμουν πολύ προσεκτικό στην τρομοθέτησή μου, γιατί όταν ο Γερμανός υπουργό είπε κάτι που είπατε κι εσείς, ε, έγινε χαμός. Έγινε πραγματικά χαμός. πώς κάνουμε τις, χαμηλότερες, τις ε, ε, κοινωνικές τάξεις με χαμηλότερο εισόδημα τις υποχρεώνουμε να φάνε αλογίσιο κρέας. Από τη στιγμή όμως που θα υπάρχει ε, σωστή ετικετοθεσία δεν υπάρχει πρόβλημα ε, να ε, διανέμεται αυτό το κρέας ε, σε όποιον θέλει να το φάει αρκεί να, το, να ξέρει τι τρώει και να μην νομίζει ότι τρώει κάτι άλλο οπότε ήμουν πάρα πολύ προσεκτικός σε αυτά που είπα αλλά παράλληλα ε, δεν ήμουν και εντελώ. δεν, δεν, δεν τήρησα σιγή ως προς το θέμα αυτό όσον αφορά τώρα τα ηνοπνευματώδη. Yes, um, αναφορά... Ερχόμουν τώρα στα πνευματόδι, έλεγα. Θα έρθει κάποιος από τη Γενική Διεύθυνση ε, ΣΑΝΚΟ. Ζητώ συγγνώμη που δεν σας δηλώσαμε την προθυμία μας να έρθουμε. Παρόλο που επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στο κάπνισμα και είναι πιο εύκολος ο στόχος από ότι το ενόπνευμα. Α, για να σας πω και γιατί το πρόβλημα στο ενόπνευμα είναι η κατάχρηση. Ενώ στο κάπνισμα ακόμα και το πρώτο τσιγάρο βλάπτει. Αλλά δεν θα πρέπει να είμαστε συγκαταβατικοί ε, με το ενόπνευμα και να λέμε ότι επειδή είναι επικίνδυνη μόνο η κατάχρηση ενοπνεύματος, ας αφήσουμε το ενόπνευμα και να ασχοληθούμε μόνο με τον καπνό. Ε, έχουμε μια στρατηγική αν θα εκπαιδεύσει θα το ξαναδούμε και όταν. Τώρα για τις τιμές. Έχουν δείξει οι μελέτες ότι για διάφορα θέματα τα οικονομικά μέτρα είναι εκείνα που αποδίδουν περισσότερο. Ορισμένοι μου λέγουν ότι οι εκστρατείε ενημέρωσης αποδίδουν καλύτερα. Δεν είναι μόνο αυτό. Αυτή τη στιγμή αυξηθεί η τιμή, συνήθως πέφτει η κατανάλωση σε όλα τα προϊόντα και στο κάπνισμα. Σε ορισμένες χώρες ακόμα και τα πατατάκια έχουν ακριβήνει γιατί ε, βλάπτουν την υγεία, γιατί παχαίνουν. Αν με ρωτάτε, ε, εγώ είμαι υπέρ τη ελάχιστη τιμή, να υπάρχει μια κατώτατη τιμή, αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα προϊόντα καπνού και αν αυτό συνάδει με το πνεύμα της εσωτερικής αγοράς και την ίδια τη συνθήκη. Δεν μπορώ να σας δώσω εδώ άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διότι δεν έχουμε κοινή θέση. Σας λέγω την προσωπική μου άποψη. Um, uh, Μάλιστα. Ε, ο κύριος Σταγιάννη δεν ξέρω αν έχει έρθει ήδη, αλλά μπορούμε να χωρέσουμε άλλες τέσσερις ερωτήσεις γρήγορα, γρήγορα. Κορέα Ντεκάμπος και άλλοι δύο ε, γρήγορα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια απευθυνάμεση ερώτηση επί τρία-τέσσερα χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχούσε και το Κοινοβούλιο το ίδιο με την οδηγία για την διασυνοριακή υγεία. Η οδηγία αυτή εγκρίθηκε πριν από δύο χρόνια. Όμως χρειάζονται και πρακτικά μέτρα ώστε κάποια στιγμή ε, από την σκοπιά της ενιαίας αγοράς να εφαρμοστεί, να είναι αποτελεσματική. Δεν ξαναμιλήσαμε για την οδηγία αυτή. Το καθόλου νέα θα πει καλά νέα ή άσχημες ειδήσει τελικά. Ευχαριστούμε. Η πιο σύντομη ερώτηση για σήμερα το απόγευμα. Εσείς πρέπει να τα πάτε καλύτερα. Κυρία Μπέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία, πολύ σύντομα, όμως σας διαβεβαιώ, για το θέμα του κανονισμού για τις ιατρικές συσκευές και τι ιατρικές συσκευέ για τη διάγνωση in vitro. Είμαι εισηγήτρια εγώ σε αυτή την επιτροπή για το θέμα αυτό και θέλω να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που κατέληξε ω τώρα σε ένα κείμενο μεγάλη ποιότητα. Όμω, η εμπορία των υψηλού κινδύνου ιατρικών συσκευών κανέναν μάλλον δεν φέρεται να ευχαριστεί ούτε το μηχανικό κλάδο, ούτε τι ενώσει ασθενών και μοιάζει για κάποιες ιατρικές συσκευές υψηλού κινδύνου με καινοτόμο χαρακτήρα η μόνη ειδική γνώση των ε, φορέων που έχουν ε, αναλάβει την έγκριση να μην είναι αρκετό αυτό. Τι προσέγγιση θα ακολουθήσουμε λοιπόν. Πρέπει να υπάρχει μια αξιολόγηση συλλογικότερη και τελείως ανεξάρτητη. Κάτι ακόμη για το ίδιο κείμενο για τις ουδέτερες δοκιμές διάγνωσης. Δεν εμφανίζονται στο κείμενο, δεν καλύπτονται, δεν θα έπρεπε όμως να συμπεριλαμβάνονται κατά τη γνώμη σας. Διότι και εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα πρόβλημα που μπορεί να είναι μείζονος σημασία για το μέλλον. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Αλλά ο Επίτροπος πρέπει να φύγει, έτσι. Το πήρε το μήνυμά σας. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Σάντεμόζε την ευκαιρία για μια πολύ γρήγορη ερώτηση. Με συγχωρείτε κύριε Μπερά, αλλά δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μου δίνετε το χρόνο. Απλώς να σχολιάσω και να πω ευχαριστώ που ήρθατε. Ευχαριστούμε που μα παρουσιάσετε το δέσμο μέτρων για την προστασία των καταναλωτών. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να ολοκληρωθεί η πρόταση πριν το τέλο τη θητεία. Είναι πολύ σημαντικό και την περασμένη μόλι εβδομάδα καθορίσαμε ένα πρόγραμμα για τη δουλειά μα. Νομίζουμε λοιπόν ότι ναι, γίνεται να ολοκληρωθεί η πρόταση πριν το τέλο τη ε, θητεία. Αυτό το μήνυμα ήθελα να στείλω. Είχα πάρα πολλέ ερωτήσει, αλλά δεν έχω χρόνο. Κρίμα. Ένα σχόλιο μόνο. Κύριε Ντεκάμπο, καμιά φορά η ανυπαρξία ειδήσεων είναι καλή είδηση. Ναι, βεβαίω και μα απασχολεί αυτό σε βάθο. 25 Οκτωβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία όταν θα τεθεί σε ισχύ η οδηγία αυτή για τη διασυνοριακή υγεία. Ήδη ε, κοιτάμε τη συγκριτική αξιολόγηση έτσι ώστε όταν τεθεί σε ισχύ ε, που θα υπάρξουν στην αρχή κάποιες παιδικές ασθένειες να φροντίσουμε να τις αντιμετωπίσουμε από την αρχή ε, πριν τις βγούμε μπροστά μας αργότερα. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι συνήθως ο κόσμος θέλει να νοσηλεύεται στη χώρα του, τουλάχιστον στη δική μου χώρα, γιατί είναι γύρω οι ασθενείς, η οικογένεια, δεν θέλει κανείς να ξενιτευτεί για να νοσηλευτεί. Ταυτόχρονα γίνεται και μια εκστρατεία ενημερωτική, όσο και διαφημιστική, ε, για τα δικαιώματα που έχουν οι ασθενείς εκτός ε, των συνόρων τους και αυτό είναι και μια συλλογή, ένα συμπίλημα της νομολογίας θέλησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τα συλλέξει όλα αυτά. Θα πρέπει να επαγρυπνούμε για την οδηγία αυτή, διότι είμαι βέβαιος ότι κάποιες κυβερνήσεις θα αποπειραθούν να δυσκολέψουν ε, αυτή την προέγκριση ή το να ζητάει κανείς προέγκριση για να μεταβαίνει στο εξωτερικό ή να τους επιβάλλουν προέγκριση όταν δεν χρειάζεται ή να βάλουν δυσκολίες ε, για το τι ε, θα τους επιστρέφουν τα ταμεία, γιατί ένας Βέλγος που πάει να νοσηλευτεί στη Γερμανία έχει επιστροφή ε, από το Βέλγικο Ταμείο τη Βέλγικη τιμή και όχι τη Γερμανική. Ε, σίγουρα αυτό θα συζητηθεί στο Βίλνιου στην επόμενη άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Υγείας. Και η Προεδρία θα ασχοληθεί και η Λιθιονική με αυτό το θέμα ποιος είναι ο στόχος 25 Οκτωβρίου να είναι άλλη μια συνηθισμένη ημέρα και όχι μια ημέρα κρίσης για την οδηγία αυτή που καλύπτει και άλλους τομείς αλλά αυτός είναι ο βασικότερος ε, να μπορεί κάθε ασθενής ατομικά να έχει τη δυνατότητα να νοσηλεύεται στο εξωτερικό. Με καμιά φορά χρειάζεται προέγκριση, ε, αλλά τελικά ε, τα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας του τον αποζημιώνουν. Κυρία Μπερά. Έχουν γίνει κάποιες προτάσεις από την Επιτροπή για ε, τα, τις ιατρικές συσκευές και το μη ιατρικό τμήμα. Με ενημερώνουν οι υπηρεσίες μου ότι επίκειται μάλλον συμβιβασμός που θα ικανοποιήσει και την Επιτροπή σας και τη Γενική Διεύθυνση Υγιεινής. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Α, για την ασφάλεια των προϊόντων ρωτήσατε. Ελπίζω η νομοθεσία αυτή να περάσει από το παρόν κοινοβόλιο κατά τη διάρκεια του της θετίας. Αλλά ξέρω, το έχω παρακολουθήσει και στο παρελθόν. Για σας 26 Μαΐου είναι η καταληκτική ημερομηνία του 2000. 14 και τους προηγούμενους μήνες μάλλον θα επιβραδυνθεί λίγο, θα είναι στο ραλαντή η λειτουργία του Κοινοβουλίου. Λοιπόν, ό,τι περάσει τους επόμενους 7 μήνες θα είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε αυτό το τομέα. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. I'm sorry I had to rush. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη που σας πίεσα, αλλά νομίζω πολλά είπαμε και πολλά σημειώσαμε. Ρεκόρ ερωτήσεων. Ξέρω ότι πρέπει να φύγετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με χαρά για πρώτη φορά σας είχαμε ενώπιό μας και με χαρά σας ξαναδούμε πολύ σύντομα. Να σας ενημερώσω ότι ο κύριος Ταϊάννη απαντά σε ερωτήσεις στην Υποεπιτροπή Άμυνας ε, για τις προμήθειες ε, άμυνας ε, και εκείνοι δυστυχώς καθυστέρησαν. Θα έρθει το συντομότερο δυνατόν. Δείξτε λίγη υπομονή. Uh, uh, Συνάδελφοι, ο κύριος Σταγιάννη έφτασε. Σας παρακαλώ να καθίσετε. Ε, μπορούμε να αρχίσουμε να δεχόμαστε ονόματα για τον κατάλογο γορτών. Φαντάζομαι, οι συντονιστές θα θέλουν να μιλήσουν. Η κυρία Ρότεβα, η κυρία Κορατσαμπίλτ, προφανώς δεν έχει φύγει κανείς ακόμα. Προτείνω, εάν συμφωνούν οι συντονιστές, διότι τρεις τουλάχιστον εδώ, να κλέψουμε λίγο το χρόνο των συντονιστών. Μπορούμε να τελειώσουμε τη συνάντηση των συντονιστών σε λιγότερο από μια μισή ώρα. Κερδίζουμε 40 λεπτά. Κύριο Κέπχαρτ, ο κύριο Βάμπ, φαντάζομαι θέλουν να μιλήσουν. Κυρία Κέπχαρτ, ο κύριο Βάμπ θέλουν να μιλήσουν, φαντάζομαι. Είναι χαρά μα να καλωσορίζουμε εδώ τον Αντώνιο Ταγιάννη. Έχουμε μια σειρά από ενδιαφέροντες προτάσεις, από ενδιαφέρουσες προτάσεις που συζητάμε. Ιδίω με την ενιαία αγορά και την ενιαία αγορά για τα αγαθά, την εποπτεία της αγοράς και μια σειρά από άλλα σχέδια. Τον, εξοπλισμό, τον ραδιοφωνικό εξοπλισμό, τα οχήματα, του κ. Μάντερς, γνωμοδότηση για λογαριασμό τη Επιτροπής Βιομηχανία για τα αρχήματα και τη στατική του 2020. Είναι πολλά τα σχέδια. Γι' αυτό κύριε Επίτροπε, ενημερώστε, μα μας και εσείς για τι δικέ σας προθέσει. Για τη σειρά από τι συναντήσει που μα περιμένουν μέχρι το τέλο αυτή τη θητεία. Οι συνάδελφοι θα έχουν και ενδιαφέρουσε ερωτήσει. Σίγουρα όμως όχι τόσο προκλητικές όσο αυτές που είχατε από την Επιτροπή Άμυνας. Και η κυρία Βάιλα, η συγγέντρια για το ραδιοφωνικό εξοπλισμό. Είναι χαρά μου να σας δώσω το λόγο. Ευχαριστώ αγαπητέ μου πρόεδρε. Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση, αλλά με κράτησαν στην δύσκολη και περίπλοκη συζήτηση στην Επιτροπή Άμυνας γιατί ε, είδαμε την ανακοίνωση που θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πολιτική αμυντικής, για την ε, βιομηχανία αμυντικής πολιτικής. Ήμουν σε άλλη αίθουσα του Κοινοβουλίου τέλο πάντων και περνάω μέσα στην ουσία. Ε, πρόεδρε, ε, πάντα για μένα είναι χαρά να έρχομαι σε αυτή την Επιτροπή, γιατί όπως ακούσατε και από τον Επίτροπο Board, για την ασφάλεια των προϊόντων και την εποπτεία της αγοράς θα δώσω και εγώ κάποια συμπληρωματικά στοιχεία. Η πρόταση υποβλήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου και ο βασικός άξονας είναι να υπάρχει ασφάλεια για τους καταναλωτές που κατά κύριο λόγο ενδιαφέρει η πρόταση αυτή. Η εσωτερική αγορά και η οικονομία μας θα λάβουν νέα τόνωση προς όφελος των επιχειρήσεων και των ε, πολιτών. Βεβαίω, είναι πολλά τα προϊόντα που δεν είναι ακόμη ασφαλή. Το 2011 το Ευρωπαϊκό Σύστημα Γρήγορη Έγκαιρη ε, Ειδοποίηση κατέγραψε. επι... κινητοποιήθηκε πολλές φορές για να ε, επισημάνει επικίνδυνες περιπτώσεις. Το 27% αφορούσε τον κλωστοφοντολογικό τομέα, το 21% τα παιχνίδια, το 11% τα οχήματα με κινητήρα, το 8% τον ε, οικιακό εξοπλισμό και το 7% τα καλλιντικά. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε για την υγεία των καταναλωτών μα να μην είναι επικίνδυνα τα προϊόντα. Η προστασία της υγείας, η προστασία των επιχειρήσεων, αλλά και η καταπολέμηση της εγκληματικής δράσης, διότι πολλές φορές η πώληση αυτών των προϊόντων ε, είναι στα χέρια του υποκόσμου. Είτε της ε, ευρωπαϊκής είτε ευρωπαϊκών εγκληματικών ομάδων, είτε εξωευρωπαϊκών. Εδώ χρειάζεται λοιπόν αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε πολλέ πρωτοβουλίε, φάσμα ευρωπαϊκής, σε Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της παραχάραξης και της νοθείας. Θέλαμε να εξηγήσουμε στους πολίτες ποιες, ποιοι είναι κίνδυνοι όταν αγοράζουν ένα παραποιημένο προϊόν. Δεύτερη πρόταση κανονισμού, αυτή που αφορά την εποπτεία της αγοράς. Το πεδίο εφαρμογής είναι ευρύτατο, διότι αφορά όχι μόνο τα καταναλωτικά προϊόντα, αλλά και τα αγαθά Επαγγελματική χρήση με εναρμονισμένε προδιαγραφέ. Και εδώ θελήσαμε να πλουστεύσουμε την ισχύουσα αρμοθεσία διότι η εποπτεία διέπεται από πολλά αριθμιστικά κείμενα σήμερα. Γι' αυτό το λόγο η πρότασή μα προβλέπει ένα ενιαίο κείμενο το οποίο θα ρυθμίζει το σχετικό τομέα. Ο στόχο είναι να υπάρχει μεγαλύτερη και καλύτερη συνεργασία των αρχών εποπτείας λόγου χάρη μέσω τη ενίσχυση, τη Τράπεζα Δεδομένων ICSMS που θα επιτρέπει την καθημερινή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων ε, αρμόδιων αρχών, ιδίω για τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων ελέγχου. Επιπλέον, θα δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό φόρουμ για την εποπτεία τη αγορά, στο οποίο θα συμμετέχουν οι αρμόδιε αρχέ των κρατών μελών, αλλά που θα προσκαλούνται και οι εκπρόσωποι ενώσεων καταναλωτών και ενώσεων επιχειρήσεων. Σε αυτό το πακέτο τη δέσμη μέτρων, πρόταση κανονισμού για την εκλασιμότητα των προϊόντων και εποπτεία της αγοράς. Αυτά τα δύο συνοδεύονται από ένα πρόγραμμα δράσης με 20 συγκεκριμένε άμεσες δράσεις για να γίνει ασφαλέστερη αγορά αγαθών για τους καταναλωτές. Για παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε τις δοκιμές ασφαλείας που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε ένα κράτος μέλος. Ε, αυτές θα εξάγονται και σε άλλα κράτη-μέλη χωρίς να χρειάζεται να επαναληφθούν. Εδώ θα αναπτυχθούν κριτήρια για τον καθορισμό τη πραγματική αποτελεσματικότητα των διαφορών συστημάτων ελέγχου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε πού απαιτείται να παρέμβουμε για να γίνει πιο ε, σταθερή η εποπτεία στην Ευρώπη. Επίση, θα αναπτυχθούν συγκεκριμένε μεθοδολογίε για να πραγματοποιούνται έλεγχοι σε αγαθά ε, υψηλή τεχνολογία και καινοτόμα προϊόντα, εφόσον έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία δύσκολα αξιολογούνται κάποιε φορέ. Εύχομαι λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει προτάσεις από τη δική σας ε, επιτροπή με νέες ιδέες και είμαι στη διάθεση της κυρίας Πιτικάιναν και της κυρίας Άλντε Μόζε για να συνεργαστούμε όσο δυνατόν αρμονικότερα. Η επανεξέταση της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά και τα βιομηχανικά προϊόντα, μια από τις βασικές προτεραιότητες στο τέλος της θητείας μας. Αυτή η επανεξέταση ε, γράφεται στη Γενική Προσπάθεια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απλουστεύσει και να ενημερώσει τι ισχύουσε προδιαγραφέ στον ε, χώρο των βιομηχανικών προϊόντων. Στην ανακοίνωση για τα βιομηχανικά προϊόντα δώσαμε στην ανάγκη να προβλέπετε ένα τεστ, μια δοκιμή ανταγωνιστικότητα, αλλά και να προχωρήσουμε σε ένα έλεγχο υγεία τη ισχύουσα νομοθεσία μέσω τη ανάλυση του σωρευτικού τύπου που έχει η υλοποίησή τη. Σε αυτό το πλαίσιο η δουλειά μας βασίζεται σε απαιτήσει και προβλήματα που έχουν εντοπιστεί από τον βιομηχανικό κλάδο, του καταναλωτέ και άλλες οργανώσεις που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών. Οι δημόσιες διαβουλεύσεις ολοκληρώθηκαν στις 17 Απριλίου και τώρα εξετάζουμε τις σχετικές ε, απαντήσεις. Ταυτόχρονα προχωρούμε στην αξιολόγηση του κεκτημένου στον τομέα των βιομηχανικών προϊόντων, όπου τα πρώτα αποτελέσματα θα γνωστοποιηθούν στα τέλη Ιουνίου του τρέχοντο έτου. Η έγκριση τη πρόταση προβλέπεται για μετά το καλοκαίρι. Άλλο θέμα ιδιαίτερη σημασία, αυτό της ε, τυποποίηση, Κάτι που είναι ακρογωνίως λήθος στην οικοδόμηση της ενιαίας αγοράς. Και ευχαριστώ την δική σας Επιτροπή για τη δουλειά που έχει κάνει σε πλήρη συντονισμό με τις δικές μας υπηρεσίες, ώστε να καταλήξουμε σε σημαντικότατες προδιαγραφές για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως προβλέπεται από το κανονιστικό κείμενο, αυτό το οποίο από κοινού εγκρίναμε, θα εργαστούμε για να ετοιμάσουμε ένα ετήσιο πρόγραμμα τη Ένωση για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση. Εδώ υπάρχουν δύο πρωταρχικοί στόχοι. Πρώτον, να ενισχυθεί η διαφάνεια σε σχέση με τι της τυποποίηση και έπειτα να εντοπίσουμε τι στρατηγικέ προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Τυποποίηση λόγου χάρη, με ένα πρόγραμμα εργασιών που θα διασυνδέει τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τυποποίηση με τη στρατηγική για την επιμηχανική πολιτική και του έξι τομεί παρέμβαση κατά προτεραιότητα, ε, όπως έχουν εντοπιστεί θα πρέπει να εγκριθεί το ετήσιο πρόγραμμα πριν από την θερινή διακοπή και αυτό υπό τη μορφή ανακοίνωση τη Επιτροπή. Δύο συγκεκριμένα παραδείγματα τυποποίηση που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών και τα οποία επεξεργαστήκαμε πρόσφατα. Ο κοινό ε, φορτιστής εδώ έχω, πρέπει να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το μνημόνιο κατανόηση για τον κοινό φροντιστήριο, όπω ετοιμάστηκε, αλλά η αξιολόγηση των υπηρεσιών τη Γενική μου Διεύθυνση στη συνεργασία με όσου συμπέραψαν το μνημόνιο κατανόηση, πρέπει να πούμε ότι ήταν θετική. Ε, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν το 90% των νέων μοντέλων κινητών τηλεφώνων που έχουν κυκλοφορήσει στην ευρωπαϊκή αγορά πέρυσι από την πλευρά των ε, όσων συνήψαν τη συμφωνία και των κατασκευαστών μπορούν να φορτίζονται με αυτό την κοινή μέθοδο. Αυτό λοιπόν είναι ένα ευχάριστο νέο. Επειδή όμως θα εκπνεύσει το μνημόνιο κατανόηση στα τέλη του 2000 εξέπνευσε μάλλον το 2012, ζητήσαμε από τους ε, ε, από όσους συμφώνησαν σε αυτό το κοινό σύστημα μία παράταση Παρά τις προσπάθειές μας δεν υπήρξε θελούσια συμφωνία μεταξύ των όσων συνυπέραψαν τη συμφωνία για άλλους λόγους και αναζητήσαμε άλλες διεξόδους. Η Γενική Διεύθυνση λοιπόν εκπώνησε μελέτη για να αποτιμήσει τα αποτελέσματα που έχουμε αποκομίσει σήμερα και επίσης τον αντίκτυπο που προέκυψε προκειμένου να υπάρξει απαραίτητη συνέχεια σε όλη αυτή την πρωτοβουλία. Επιπλέον, την περασμένη εβδομάδα 8 παραγωγή ε, κινητών τηλεφώνων υπέγραψαν την ε, επιστολή προθέσεων που ε, δηλώνει ότι πρόκειται να προχωρήσουν με το μνημόνιο κατανόηση. Έτσι, η πίεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή του ανάγκασε να επιταχύνουν για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία μεταξύ μα και αυτό μα κάνει να ελπίζουμε. Βεβαίω, εάν δεν υπάρξει μονογραφή τη συμφωνία, δεν μπορώ να εμπιστεύομαι πλήρως την ε, μελέτη αντικτύπου. Εδώ πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αλλά θα ήταν σημαντικό να πούμε στους καταναλωτές ότι υπάρξει, θα υπάρξει παράταση της συμφωνίας που εκτός από τα κινητά τηλέφωνα θα καλύπτει και τα smartphone αλλά και τους, τις συσκευές ε, MP3 και τις ταμπλέτες και τις ε, ψηφιακές κάμερες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πράσινα οχήματα, το πρόγραμμα δράση ΚΑΤΣ 2020 που εγκρίθηκε πρόσφατα δείχνει τι κάνουμε προ αυτή την κατεύθυνση το 2010, όπω ξέρετε. Ευρωπαϊκή φορεί τυποποίηση ασχολήθηκαν με την αναμονισμένη λύση τη διαλογικότητα των φορτιστών μπαταρία για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά λόγω τη Ιταλική και καλλική ιδιαιτερότητα δεν βρέθηκε λύση. Κυρίω λόγω τη αντίσταση τη Ιταλική βιομηχανία. Οι ε, Ιταλικέ εταιρείε ήταν ε, υπέρ τη γερμανική πρόταση. Τα πράγματα ήταν περίπλοκα, αλλά τελικά καταλήξαμε σε μια πρώτη συμφωνία και στη βάση της έκθεσης της ε, ομάδας μελέτης ΕΝΣΕΝΕΛΕΚ η οποία ε, κατέληξε ότι δύο είναι οι βασικοί φορτιστές που πρέπει να χρησιμοποιηθούν από, άποψη της από την άποψη τη ασφάλεια. Έτσι, το Γενάρη φέτο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια νομοθετική πρόταση για να βεβαιώσει ότι θα υπάρξει διαλογικότητα στις, ε, στους φορτιστές μπαταριών των ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζουμε λοιπόν ότι όλη αυτή η διαδικασία θα προχωρήσει. Προχωρώ προς την Προ το συμπερασμά μου, προ την ολοκλήρωση τη ομιλία, για το e-call, την ηλεκτρονική κλίση. Εδώ, όπω ξέρετε, σε συνεργασία με την Επιτροπή σα, ασχοληθήκαμε με την εγκαθίδρυση τη υπηρεσια e e-call. Εργαζόμαστε, λαμβάνοντα υπόψη τι συστάσει του Κοινοβουλίου σχετικά, όπω εγκρίθηκαν τον περσινό Ιούνιο. Όπω θα ξέρετε, η εθελούσια προσέγγιση ήταν ε, ανεπαρκή ω τώρα. Γι' αυτό έπρεπε να εγγυηθούμε την ε, διάδοση τη υπηρεσία αυτή, τη e-call, βάσει του νούμερου, με τον αριθμό 112. Αυτό επιχειρήθηκε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έω την 1η Οκτωβρίου του 2015. Το Μάιο θα εγκρίνουμε δύο νομοθετικέ προτάσει. Έναν κανονισμό που θα καθιστά δεσμευτικό, υποχρεωτικό το σύστημα e-call στα οχήματα και έπειτα μια απόφαση που θα, οργανώ, που θα ορίζει συγκεκριμένα πρότυπα για τις εθνικές υπηρεσίες επιγόντων. Έπειτα, με τα νομοθετικά μέτρα, θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε, αφού λάβουμε υπόψη και τις απόψεις των κρατών μελών, το τι επιθυμεί αυτό η μηχανία, και τα δίκτυα των παραγωγών για να είναι αποτελεσματική η χρήση της υπηρεσίας e-call. Τώρα για τις καθυστερήσεις πληρωμών, όπως ξέρετε το περασμένο Μάρτιο εγκρίθηκε η μεταφορά της οδηγίας, πέρασε η καταληκτική ημερομηνία και για αυτό το στάδιο και πρέπει να σας πω ότι ως σήμερα ξέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μόνο 18 κράτη-μέλη έχουν κοινοποιήσει την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στην Εθνική Νομοθεσία πέραν των αστείων τώρα. Νομίζω λίγο πολύ καλά τα πήγαμε. Έχουμε οργανώσει εκστρατείε ευαισθητοποίηση σε όλα τα κράτη-μέλη. Εκεί συμμετείχαν πολίτε, εταιρείε, επιχειρήσει με σκοπό να ενημερωθούν για τους νέους ευρωπαϊκούς κανόνες. Προφανώς χώρες που προβλέπουν μικρότερη διορία για τις πληρωμές δεν χρειάζεται να την παρατείνουν. Απλώς όριο είναι οι 30 μέρες και κανείς δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Κάθε χώρα έχει τα δική τη ομοθεσία που μπορεί να ορίζει να γίνει πληρωμή σε 10 μέρες. Αυτό συνάδει πλήρω με τόσο ορίζει οδηγία. Απλώ ο στόχο είναι να μην ξεπερνιέται το όριο των 30 ημερών, που είναι το μέγιστο όριο. Αυτό ήταν το πνεύμα του νομοθέτη. Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε το βασικό όριο και εδώ στόχο ήταν να βοηθήσουμε τι επιχειρήσει. Εάν σε μια χώρα λοιπόν οι κανόνε διαφέρουν και είναι και καλύτεροι, αφού ακολουθούν το πνεύμα τη οδηγία, δεν χρειάζεται να αλλάξει τίποτα. Δεν χρειάζεται να υπάρξει επιπλέον καθυστέρηση. Εμείς θα φροντίσουμε η οδηγία να γίνει σεβαστή και να εφαρμοστεί ορθώς σε όλη την επικράτεια της Ένωσης και θα προσπαθήσουμε, όπως ε, ξεκίνησε ήδη να γίνεται σε κάποια κάτι μέλη, ιδίω στη δική μου χώρα προέλευσης, γιατί εκεί υπήρχε μεγαλύτερη καθυστέρηση, θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε λοιπόν μαζί με τις μελλοντικέ ε, οφειλές να πληρωθούν κάποιες και αναδρομικά. Δεν μπορούμε να καταδικάσουμε τις επιχειρήσεις σε θάνατο λόγω χρεών των δημοσιοδικήσεων. Όχι. Και το δημόσιο, όπως έχει την, ε, το δικαίωμα να απαιτεί από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να πληρώνουν φόρους, πρέπει και εκείνοι να πληρώνουν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος όσα οφείλουν στους ιδιώτες και τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για πολλά ζητήματα που θέσατε. Έχουμε σίγουρα ερωτήσεις. Να σας πω. Ποιοι είναι. Σφαμπ, Κέπχαρτ, Ρούλε. Μετά. Ρόιτα, Κοράτσα Μπίλτ και Άριας. Μετά Βάλερ και Κανιέτσι. Και μετά η κυρία Λεγκρίπ. Υπάρχει κανένας άλλος. Right, so I think we have sort of three batches then, so we'll do them in threes. Λοιπόν, Σφαμπ, Γκέμπχαρτ, Ρούλε. Παρακαλώ να είστε σύντομοι, ώστε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας ε, όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ώρα που είχαμε προβλέψει. Κύριε Σφαμπ. Πρόεδρε, πάντα προσπαθώ να είμαι ευσύνοπτος. Ευχαριστώ κύριε Πίτροπε, χαίρομαι για την παρουσία σας. Ε, για τα αυτοκίνητα για τις ενιαίες πινακίδες κυκλοφορίας είναι πάρα πολύ χρήσιμη πρόταση για τους πολίτες καταναλωτές που καθημερινά κυκλοφορούν στην Ευρώπη και διασχίζουν σύνορα. Ε, θέλω να ρωτήσω όμως κάτι άλλο για θέματα που χρονίζουν λίγο. Θέλουμε να κάνουμε μια ερώτηση ε, για το εξής θέμα. Στη Γερμανία, βάσει της οδηγίας για τις καθυστερημένες πληρωμές, χρειάζεται αλλαγή ε, της ένομης τάξης Γερμανίας, λέγουν ορισμένοι. Εγώ θεωρώ ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά ο αρμόδιος επίτροπος θα πρέπει γραπτός να το επιβεβαιώσει για να μπορέσουν να το καταλάβουν και να λάβουν γνώση και οι υπουργοί στο Βερολίνο. Και θα παρακαλούσα να μας απαντήσετε σήμερα προφορικά. Και αποφασίσαμε πρόσφατα την οδηγία για τα οικοδομικά υλικά και υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις ε, τελικές που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο κατασκευαστικός κλάδος. Η οικοδομή γενικότερα περιμένει απάντηση. Μπορείτε να μας απαντήσετε. Ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, Mrs. Ευχαριστώ κυρία Γκέπχαρτ. Ευχαριστώ κύριε Ταγιάννη για τα σαφή σας λόγια και πάλι για αυτά που είπατε ότι δεν πρέπει να αλλάξει η γερμανική νομοθεσία για ε, τις καθυστερημένες πληρωμές και χρειάζεται κάποια παράταση. Το εξηγήσετε πολύ ωραία. Υποστηρίζω πολύ τους αυτά που είπε ο κύριο Σβάπ. Μπορείτε να τα πείτε και στου υπουργού μα στο Βερολίνο ή να του τα γράψετε για να τα χωνέψουν κι αυτοί. Διότι είναι μια ανήρη ιστορία αυτή και μια συζήτηση ανίποτη. Και πάλι κατηγορείται η Ευρώπη για κάτι για το οποίο δεν φταίει. Και δημιουργεί αυτό και μεγάλη δυσφορία στις επιχειρήσεις όπου καθυστερούνται οι πληρωμές. Ε, θα ήθελα να σας συγχαρώ επίσης για τη διαλειτουργικότητα των φορτιστών, των ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών. Αυτό είναι πραγματικά κάτι που βοηθάει πάρα πολύ τους καταναλωτές. Συνεχίστε σε αυτή την ε, κατεύθυνση και επίσης το δέχονται πάρα πολύ θετικά. Και δεν είναι μόνο καλό για τους καταναλωτές, για το περιβάλλον και γενικότερα γιατί πραγματικά θα εξοικονομήσει πολλά χρήματα. Ε, να πω δύο λόγια για την βιομηχανική πολιτική. Έκανα ε, πρόσφατα την γνωμοδότηση, την κάνω αυτό το καιρό και θα ψηφίσουμε αύριο. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω και εσάς που φέρατε την πρόταση, διότι η κρίση που ζούμε σήμερα δείχνει ότι Φύγονται περισσότερο τα κράτη από την κρίση που έχουν επικεντρωθεί στις υπηρεσίες και όπου έχουμε ένα υγιές μείγμα ανάμεσα στη βιομηχανική παραγωγικότητα και στην παραγωγικότητα των υπηρεσιών είναι καλύτερη η κατάσταση και ε, αντέχουν περισσότερο στην κρίση. Αυτό νομίζω πρέπει να μας απασχολήσει πιο πολύ και να δραστηριοποιηθούμε. Ευχαριστώ. Now, I think uh, ε, κυρία Ρούλα. Οι ερωτήσεις μου έχουν ήδη τεθεί καλύφθηκα. Ε, μία παράκληση για τα προϊόντα, για τα οικοδομικά προϊόντα και υλικά. Το είπε και ο κύριος ε, Σφάπ για τις κατεξουδότηση πράξης ε, να περάσει το συντομότερο για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε την πρόταση και να λυθεί αυτό το θέμα της νομικής ασάφειας που επικρατεί αυτόν τον καιρό. Uh, ο κύριος Δεγιώνας ε, προσταθεί αργότερα στον κατάλογο ομιλητών, αλλά αν χρειαστεί θα του δώσουμε και πραγωγή. Επίτροπε, θέλετε να απαντήσετε σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις πληρωμών. Οι δύο ερωτήσει ε, του κυρίου Σφάμπ και της κυρίας Κέπχαρτ θα μπορούσαν να απαντηθούν απλούστατα και με Εάν η Γερμανία έχει κανόνες που προβλέπουν ότι η πληρωμή πρέπει να γίνεται σε χαμηλότερη διορία, σε μικρότερη διορία από τις 30 ημέρες, ε, δεν χρειάζεται η Γερμανία να τις αλλάξει κατά την άποψή μου. Εάν υπάρχουν συγκεκριμένες ε, εξαιρέσεις θα το κοιτάξω, αλλά από άποψη τεχνική και νομική αυτή είναι η κατανόησή μου και η ερμηνεία μου. Είναι ανώτατο το όριο. Εάν θέλει μια χώρα πληρώνει γρηγορότερα, θα παραβιάσετε τι οδηγίε, Θα ήταν να μου λέτε ότι η Γερμανία πρέπει να πληρώσει σε 40 μέρε. Αυτό θα ήταν παραβίαση της οδηγία. Τώρα, η οδηγία πρέπει να γίνεται σεβαστή και στα υπόλοιπα τμήματά τη. Για αυτά που είπε ο κύριο Φαμπ, το συζητήσαμε και η κυρία Γκέφα, το θυμάται. Ε, αλλά για τη διορία. Εάν μια χώρα προβλέπει διάστημα μικρότερη διάρκεια, το σημαντικό είναι να εφαρμόζεται και το υπόλοιπο τη οδηγία. Εάν όμω ένα βουλευτή ο κύριο Φάμπε, κυρία Γκέμπχαρτ ε, ε, υποβάλλουν άμεση ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα λάβετε και απάντηση. Εγώ θα φροντίσω να το ελέγξω, να το παληθεύσω και με την νομική μα υπηρεσία, ώστε να εξηγηθεί με απόλυτη σαφήνεια ότι η Ομοσπονδιακή Ομοσπονδιακή ε, Δημοκρατία της Γερμανίας μπορεί να μεταφέρει την οδηγία με τον ένα τον άλλο τρόπο. Αλλά ήδη σα καθησυχάζω με το που θα γυρίσω στο γραφείο μου θα ζητήσω από τι υπηρεσίε τη Γενική Διεύθυνση να μιλήσει με το αρμόδιο Υπουργείο τη Ομοσπονδιακή Γερμανία τη Γερμανία για να αποφευχθεί κάθε πρόβλημα και να μην υπάρξει καμία περαιτέρω διαφιλονικία. Το συζήτησα όμω και πριν έρθω εδώ με τον Γενικό μα Διευθυντή. Είπε η υπόλοιπη Ευρώπη, άλλες χώρες. Όταν πήγα στη Φιλανδία, ο πρόεδρος ε, του βιομηχανικού συνδέσμου μου είπε ότι είμαι πάρα πολύ, παίρνω χαλαρά μέτρα, διότι πρέπει να αφήνω τις εταιρείε να πληρώνουν πολύ αργά. Οι φιλανδικές εταιρείε πληρώνουν σε 10-15 μέρες. Τώρα τι να σας πω, μπορεί να κάποιος να θέλει και το όριο των χιλίων ημερών, αλλά η φιλοσοφία του νομοθετικού κειμένου είναι να δώσει συγκεκριμένε απαντήσει. Να μην πτωχεύσουν οι επιχειρήσει εξαιτία των καθυστερήσεων πληρωμών. Εάν κάποιο θέλει να πληρώνει γρηγορότερα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, είμαστε σε απόλυτη συμφωνία. Τώρα, ω προ την υπόλοιπη εφαρμογή τη οδηγία, εντάξει, θα το δούμε από νομική πλευρά και η νομική υπηρεσία θα κάνει ό,τι δει. Όμω θα σα απαντήσω εάν υπάρξουν ε, απορίε. Τέλος πάντων σήμερα απόγευμα ήδη θα ζητήσω από τις υπηρεσίε τη Γενικής Διεύθυνσης να έρθουν σε επαφή με την κυβέρνηση τη Ομοσπονδιακή ε, δημοκρατία τη Γερμανία για να αποφευχθεί κάθε ε, παρεξήγηση. Σε ό,τι αφορά το θέμα των ε, οικοδομικών προϊόντων τη κατεξουσιοδότησης πράξη, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε όλες τις επίσημες διαδικασίες από την 1η Ιουλίου φέτος. Τότε θα έχει επισήμως ε, πια καταρτιστεί το δικαίωμα να γίνει αυτό βάσει του άρθρου 68 και θα υπάρχει σαφής ε, συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου. Αφού γίνει λοιπόν και έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπορέσουμε με τις πράξεις αυτές ε, να προχωρήσουμε και στη θέση ισχύ το φθινόπωρο φέτος. Θα εργαστούμε λοιπόν μαζί. Από την 1η Ιουλίου πάντως θα ξεκινήσουν και τα επίσημα βήματα της διαδικασίας. Uh, Ευχαριστώ. Επόμενοι ομιλητές και θα σας παρακαλέσω και πάλι να είστε σύντομοι και ε, είναι η κυρία Ρόιτοβα, η κυρία Κοράτσα Μπίλ και ο κύριος Αρίας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για όσα μας είπε. Θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι πολύ με τον τρόπο διαπραγμάτευσης των, ε, του πακέτου 9 οδηγιών ε, με ε, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Προεδρία. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που είναι λιγότερο σημαντικό για την κατάργηση της θερινής ώρας. Υπάρχει μια πρωτοβουλία των πολιτών στην Τσεχία. Προσπαθούμε να μαζέψουμε ένα εκατομμύριο υπογραφές σε διάφορα κράτη-μέλη. Η απάντηση ήταν ότι δεν ήταν ένα αρκετά σημαντικό ζήτημα. Είναι όμως κάτι το οποίο πραγματικά δημιουργεί πρόβλημα στον κόσμο. για λόγους όπως ε, κατανάλωση ενέργειας κλπ. Με ρωτούν τα μέσα μαζική ενημέρωση, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εσάς, έχετε σκοπό να εμβαθύνετε σε αυτό το θέμα. Γιατί σε πολλούς πολιτικούς φαίνεται να είναι ένα τίποτα, αλλά πραγματικά ενοχλεί του Ευρωπαίους πολίτες και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συνεργαστεί μαζί μα δεν μπορούμε τίποτε να κάνουμε. Πώς το συνδέεται αυτό με τον κύριο Ταγιάννη, ότι ευθύνεται και για τη θερινή ώρα. Μπράβο, πώς τα καταφέρατε αυτά. Δεν ξέρω. Ε, κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόταση για την εποπτεία της αγοράς. Ε, για τις καθυστερημένες πληρωμές, επειδή είναι δικό σας προϊόν, για το B2B, business to business. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μεταγράψει αυτό σε πρόταση, αλλά θέλουμε τώρα να μην υπάρχει πλέον ελευθερία σύναψη σύμβαση. Το B2B δηλαδή να, να περιορίζεται σε 30 μέρες υποχρεωτικά. για τις μικρές εταιρείες αυτό δεν είναι εφικτό. Για παράδειγμα, εστιατόρια, ξενοδοχεία, ε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα επηρεαστούν πολύ. Δεν θα πρέπει να υποχρεούνται να, πληρώνονται, να πληρώνουν όταν υπάρχει έλλειψη ροής κεφαλαίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς να μας πείτε πώς πιστεύετε ότι το πνεύμα του ό,τι αποφασίσαμε εδώ, του ότι έγιναμε εδώ και αυτό το οποίο τώρα η ε, αντιπολίτευση στη Σουηδία ε, προσπαθεί να υπονομεύσει, ε, ποια είναι η δική σας άποψη για το θέμα της ασφάλειας των προϊόντων. Μία διευκρίνηση για την ε, ε, ένδειξη προέλευσης. Οι καταναλωτές θέλουν περισσότερη ίχνη λασιμότητα, αλλά θα ήθελα να μου πείτε τη δική σας άποψη, γιατί ε, είναι μεγάλη η διασύνδεση, δηλαδή ε, ο σχεδιασμός γίνεται σε ένα ε, μέλος, κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραγωγή, η κατασκευή γίνεται στην Κίνα, μετά η συναρμολόγηση γίνεται αλλού και μιλάω από υφάσματα μέχρι άλλου είδους προϊόντα. Θα ήθελα να μου πείτε πώς αυτό αποτελεί προστιθέμενη αξία για τον καταναλωτή και τι γίνεται με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι επιπλέον το διοικητικό κόστος, έχετε σκοπό να το κάνετε αυτό αυτό ενδεχομένως ηλεκτρονικός, ε, ψηφιακός, μήπως μπορείτε να μας το εξηγήσετε λίγο περισσότερο, γιατί κάποια κράτη-μέλη υποστηρίζουν ότι το αποτέλεσμα θα είναι πραγματικά ένα εμπόδιο ε, στο εμπόριο. Θα ήθελα να σας συγχαρώ τέλος, γιατί βλέπω ότι την επιχειρηματικότητα των γυναικών ε, πρέπει, την υποστηρίζετε πολύ και θα έπρεπε να διαβάσετε το ψηφιακό περιοδικό, ευχαριστώ πάρα για να το διαπιστώσετε, Ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας. Ο κύριο Άρια. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Αντιπρόεδρο Ταγιάννη για την παρουσία του εδώ. Θα ήθελα να πω μόνο το εξή. Είμαι πάρα πολύ περήφανο που έχω την ευκαιρία την Παρασκευή να παρουσιάσω ε, την οδηγία για την αφαιρεγκαιότητα ε, με τον κύριο Καγέχα και τον Υπουργό Σόρια θα παρουσιάσω στην Ισπανία αυτό το θέμα. Πραγματικά πρέπει να βοηθήσουμε ε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, και είναι πολύ καλό για να μπορούν οι μικρομεσαίες να βγαίνουν από την κατάσταση που ζουν τώρα και με την καθυστέρηση των πληρωμών. Των των οχθέντων πρέπει να σας πω ότι στις μικρομεσαίες θα πρέπει να υπάρχει ισότητα ευκαιριών και ισότητα συνθήκων με τις μεγάλες εταιρείες για να μπορούν να δρουν σε έναν ανταγωνισμό ή ακόμα και με τις δημόσιες επιχειρήσεις. Οι μεγάλες εταιρείες μπορούν πιο εύκολα να αντρούν κονδύλια από το δημόσιο τομέα ή ακόμα και να συμμετέχουν σε κρατικές προμήθειες, σε διαγωνισμούς. Και τώρα με τις ψηφιακές προμήθειες μπορούν πιο εύκολα και μικρομεσαίες να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς. Και για άλλη μια φορά πραγματικά χαίρομαι που πιέζετε για ε, την ολοκλήρωση της ψηφιακής αγοράς και βοηθάτε όσο μπορείτε ε, για να ε, ενισχύει η ψηφιακή αγορά της μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να μπορούν να ευημερούν και να ανθούν. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον Επίτροπο για να απαντήσει, να σας πω ποιοι θα είναι οι τρεις τελευταίοι που θα ρωτήσουν, μην τυχόν και γραφτεί και κανένα άλλο, ε, Βάιλερ, Κανιέτε και Λεγκρίπ. Εντάξει, τέλος, λίγοι εδώ κλείνει ο κατάλογος. Να είστε έτοιμοι με σύντομες ερωτήσεις. Ε, παρακαλώ τον Επίτροπο να απαντήσει αυτές τις τρεις ερωτήσεις που μόλις ακούσαμε. Πολύ σύντομα. Πρώτη φορά ε, έχω τέτοια έτοιμα. Ε, για το ερώτημα της κυρίας Ρόιτοβα και για τη θερινή ώρα. Τώρα το θέμα που Πρώτη φορά λαμβάνω τέτοιο αίτημα και δεν έχω σκεφτεί τι θα έκανα σε αυτή την περίπτωση. Για την κυρία Κοράτσα, η Σουηδία είναι μια από τι 18 χώρε που ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την γνωστοποίηση τη μεταφορά τη οδηγία. Αυτό απάντησε στην ερώτησή σα, γιατί ενημερώσαμε τα κοινοβούλια που έχουν ήδη γνωστοποιήσει τη μεταφορά τη οδηγία ε, για τις καθυστερήσει των ε, πλεωμών ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κύπρο, Μάλτα, Ιταλία, κάτω χώρες, Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία, Βουλγαρία, Λιθουανία, Φινλανδία, Πολωνία, Σλοβενία, Γαλλία, Αυστρία, Εστονία Λουξεμβούργο και προς τιμήν του κυρίου Χάρμπουρ το στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βεβαίω τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποτιμήσει την μεταφορά αυτή καθεαυτή, αν υπήρξαν προβλήματα, εάν χρειάζονται διορθώσεις, προσαρμογέ του κειμένου, αλλά νομίζω ότι μάλλον η οδηγία έχει μεταφερθεί κατά τρόπο ορθών. Πρώτη μας πρωτοβουλία λοιπόν θα είναι να ε, ενημερώσουμε, να ζητήσουμε τι υπόλοιπες χώρες να μας πούν τι γίνεται με την μεταφορά σε κίνηση Δεν μπορεί να αλλάξει η κατεύθυνση, ο προσανατολισμός αυτός που σας ανησυχεί. Εάν υπάρχει ένας κανόνας που βελτιώνει τα πράγματα, λαμβάνεται υπόψη, αλλά εάν κάτι μεταβάλλει την οδηγία, ε, δηλαδή εάν για το B2B προβλέπεται εξαίρεση και συμφωνία και αν η συμφωνία αυτή δεν είναι επιζήμια για την μικρομεσαία επιχείρηση, αυτό θα είναι το σημείο κλειδί, τότε μπορεί να κάνει καταγγελία η μικρομεσαία επιχείρηση και να επικαλεστεί τον κανόνα που διέπει τη συμφωνία ιδιωτικού δημόσιου τομέα. Δεν μπορεί να μεταφερθεί η οδηγία αλλοιώνοντά την. Γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν θα είχε και νόημα. Όλες λοιπόν οι αξιολογήσεις νομικού χαρακτήρα θα γίνουν. Θα γίνουν και μάλιστα με προσοχή και τη δέουσα. Γιατί κάθε παραμικρή λεξούλα αξιολογείται από την νομική υπηρεσία έτσι ώστε να υπάρξει και ομοιογενής μεταφορά. Δεν μπορούμε αλλιώ να έχουμε ενία αγορά εάν δεν έχουμε και σωστή μεταφορά των οδηγιών. Δεν μπορεί να έχουμε διαφορετικέ μεταφορέ τη οδηγία από χώρα σε χώρα και οι καταναλωτέ να προστατεύονται διαφορετικά ε, αυτοί και τα δικαιώματά του από χώρα σε χώρα. Θα φροντίσουμε να σα ενημερώσουμε εφόσον υπάρξουν παρατηρήσει και από το βασίλειο της Σουηδίας για, το, για τη μεταφορά της οδηγίας. Το μελετούν αυτές τις νομικές μας υπηρεσίες. Κοιτάξαμε τι γίνεται με τη μεταφορά στην Ιταλία. Εκεί έγινε μια παρατήρηση και η Ιταλία φρόντισε να αποστείλει ερμηνευτικές εγκυκλίους ώστε να μεταφερθεί σωστά. Στη Σουηδία ακόμα βρισκόμαστε στη φάση της εξέτασης. Θα σας ενημερώσω λοιπόν εφόσον υπάρξουν προβλήματα. Κάτι ιδιαίτερο δηλαδή. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ίχνηλασιμότητα, προτείναμε ένα ε, νομοθετικό κείμενο το οποίο θα καθησύχαζε τις ανησυχίε που έχουν αφαιρεστεί σε επίπεδο ΠΟΕ ω προ το παλιότερο κείμενο της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Λασιμότητα. Η προηγούμενη πρόταση κινδύνευε να μην εξασφαλίσει επαρκές επίπεδο ανταγωνισμού, διότι υπήρχε ένα στοιχείο εχνελασιμότητας για τα εξαγόμενα προϊόντα, για τα εισαγόμενα μάλλον προϊόντα και όχι για τα ευρωπαϊκά. Η πρόταση του κανονισμού που προβάλαμε στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο προβλέπει ίχνηλασιμότητα για όλα τα προϊόντα που φτάνουν και κυκλοφορούν στην Ευρώπη και κυρίως για όσα εισάγονται στην Ευρώπη. Υπάρχει λοιπόν πλέον ίση μεταχείριση για όλα τα προϊόντα. Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα, τα κατασκευασμένα, τα επεξεργασμένα, εδώ ισχύει ο τελωνιακός κώδικας. Η τελευταία ε, εξέλιξη είναι αυτή, η τελευταία είναι μέρος μάλλον του κώδικα, είναι αυτή που ισχύει. Εάν ε, τώρα έχουμε υπόψη το σήμα Made in Europe, όπου βέβαια στο τελικό αποτέλεσμα το ύφασμα είναι κινέζικο και έχουν μπει μόνο κουμπιά ευρωπαϊκά. Εκεί δεν μπορεί να πει το σήμα Made in Europe. Εάν όμω όλο το ένδυμα λόγου χάρη έχει κατασκευαστεί στην ε, Ευρώπη και μόνο τα κουμπιά έχουν κατασκευαστεί στην Κίνα, εκεί μπορούμε να βάλουμε το Made in Europe. Πάντω, ε, αυτό που ισχύει είναι οι κανόνε του τελωνιακού κώδικα, ό,τι αφορά την αρχή. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτά που ρώτησε ο κύριος Αρίας Ετσεβερία, θα ενημερώσουμε για όλα τα σχετικά με τον ψηφιακό χώρο, διότι αυτό αφορά πάρα πολύ το μέλλον και το τι θα γίνει με τις δημόσιες προμήθειες και πώς θα διαμορφωθεί το κοπείο για τις μικρομέσες επιχειρήσεις. Όλη μας η φιλοσοφία εδώ θα είναι καθοριστική σημασία και ό,τι σκεφτούμε για τον ε, τομέα των ψηφιακών θα το κάνουμε με μεγάλη προσοχή. Δεν μπορούμε παρά να απαντήσουμε με θετικό τρόπο προς τις προτροπές του κυρίου Αρίας. Ευχαριστώ. Thank you Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα η κυρία Βάιλερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα φαντάζεστε ότι και εγώ θα επανέλθω στην οδηγία για τις καθυστερημένες πληρωμές. Είμαι και εισηγήτρια άλλωστε. Και ενδιαφέρομαι να δω εκ των υστέρων και να καταλάβω πώς θα ε, μεταφερθεί αυτό και πώς θα εφαρμόζεται πότε. Μια οδηγία που περίπου εγκρίθηκε εδώ ομόφωνα και στο Συμβούλιο οφείλω να πω, περίπου ομόφωνα με τρεις αποχές, ξαφνικά έχουμε δυσκολίες στη μεταφορά της. Με 14-15 άρθρα. Ουσιαστικά είναι μικρό το κείμενο και σαφές τις οδηγίες, προβληματίζει στην εφαρμογή του. Και για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν θα είμαι τόσο ευγενική όπως οι συνάδελφοι προαναλύσαντες. Έχω την αίσθηση ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη αυτό είναι εσκεμμένο. Τουλάχιστον στη δική μου χώρα μπορώ να θυμηθώ ότι από την αρχή ε, ήταν κατά. Στο τέλος ψήφισε αποχή η Γερμανία, αλλά θα επιθυμούσε να είχε καταψηφίσει. Και στη Γερμανική Βουλή δεν ξετρελάθηκαν. Και τώρα ε, είναι οριστικό αυτό. Και καλό θα ήταν κύριε Επίτροπε να ε, τα ξεκαθαρίσετε τα πράγματα και χαίρομαι που θέλετε να το κάνετε, αλλά είπατε ότι θα διαβιβάσετε την άποψή σας στο Γερμανό Υπουργό. Μα δεν είναι ένας, είναι οι δύο φιλελεύθεροι υπουργοί, οι οποίοι τσακώνονται και για την αρμοδιότητα. Που είναι η δικαιοσύνη και η οικονομία. Και οι δύο φιλελεύθεροι αρμόδιοι και έχουν τα πράγματα μπερδευτεί. Καλό είναι να το ξεκαθαρίσετε και για εμάς τους βουλευτές που εδώ και καιρό αντιμετωπίζουμε παρόμοια προβλήματα στην νομοθεσία. Είναι και πάλι ένα ωραίο παράδειγμα αυτό. Κάνουμε καλούς νόμους και ωραίους και μετά δεν εφαρμόζονται, δεν μεταφέρονται σωστά στην νομοθεσία μας. Είτε ανεπαρκώς, είτε εσφαλμένα, είτε δεν ξέρω τι. Ε, και το αποτέλεσμα κολλάει στις Βρυξέλλες. Γιατί αυτή τη ρετσινιά ε, ε, έχει οδηγία ότι φταίνει οι Βρυξέλλες, όχι τα κράτη-μέλη για τον τρόπο που τα μεταφέρουν και τα εφαρμόζουν. Και θα πρέπει όλοι να ανησυχούμε και να φροντίσουμε να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Αυτή η μεμψημυρία, ε, αυτές οι δυσφορίες και οι δυσάρεστες δηλώσεις από όλα τα κόμματα, γιατί έχουμε και ε, ε, εκλογές σε λίγο και θα τα φορτώσουν όλα στις Βρυξέλλες. Διάβασα μια δήλωση που κάνατε εσείς στον τύπο και παρακαλώ να το διαδώσετε. Αναφερθήκατε σε μια μελέτη που κάνατε, που αναθέσετε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μελετήθηκε η κατάσταση ως προς τις ενισχύσεις που παίρνουν από τις Βρυξέλλες. Και ήταν πολλές επικρίσεις για το REACH και τα λοιπά που είναι μεγάλα προγράμματα και έργα δύσκολα. Με το REACH πραγματικά θα έχουμε μεγάλες δυσκολίες ακόμα στο μέλλον. Αλλά ένα σημείο αναγνωρίστηκε από τις μικρομεσαίες ως το πιο σημαντικό και ως καλύτερη βελτίωση και το επένεσαν. Ήταν αυτή η οδηγία για τις πληρωμές ε, και εγώ τα μοιράζω παντού όπου μπορώ και όπου βρεθώ, αλλά σε μεγάλες και σοβαρές και πολλές εφημερίδες αυτά δεν γράφονται. Να τα πείτε αυτά σε όλους και το Κοινοβούλιο σίγουρα μέχρι τέλη του έτους θα τα παρακολουθήσει όλα αυτά για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται και μεταφέρει τη οδηγία και όχι προφόρμα για τα μάτια. Ένα δεύτερο που θέλω να φέρω είναι επίσης ε, κάποια θετικά που αναφέρατε για την εναρμόνιση των φορτιστών και των μετασχηματιστών για την ε, ε, κατανάλωση για τους καταναλωτές και εγώ στην έκθεσή μου έχω συζητήσει με τις υπηρεσίες σας ε, για τους ασυρμάτους και το ραδιοφωνικό σήμα. Έχει γίνει μια συμφωνία κυρίων υποτίθεται, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την έχει καταγγείλει και δεν ενδιαφέρεται να συνεργαστεί σε αυτή την εθελοντική συμφωνία. Και εγώ ρωτώ καλά τι του τσίμπησε, τι του έπιασε ξαφνικά, γιατί τόσο καιρό ήταν πολύ καλή η συνεργασία μα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και η ε, απάντηση ήταν ότι, α, ξέρετε, διαπιστώσαμε ότι με τους μετασχηματιστές και τους φορτιστές και άλλα ανταλλακτικά ε, από εκεί είναι το κέρδος, από εκεί βγάζουν κέρδος αυτοί που τα παράγουν κατασκευαστέ και όχι από την ίδια τη συσκευή, από τα διάφορα αξεσουάρ. Ε, και εγώ εκεί στην, στην τεχνική χρήση ε, ραδιοφωνικών σταθμών συσκευών ε, θέλω να το βάλω στην έκθεσή μου και αν δεν ε, γίνεται αυτό να ακολουθηθεί εθελοντικά, τότε να το κάνουμε δια νόμου, υποχρεωτικό. Ευχαριστώ κυρία Καμιέτε. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ε, επενέσω γιατί αρχίσατε να κάνετε επισκέψεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωση ε, φέτος. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία για να βοηθήσετε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να έχουν νέους εταίρους εκτός από ε, αυτούς που έχουν ήδη. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε σκοπό να συνεχίσετε αυτή την πρωτοβουλία στο δεύτερο τμήμα, το δεύτερο εξάμεινο του έτους και το 2014. Ίσως κάτι που θα μπορούσατε να προτείνετε είναι <laughs> μέλη της Επιτροπής μας να μπορούμε και εμείς γέρος να λαμβάνουμε ε, ενημέρωση την οποία θα μπορούμε να ε, διαβιβάζουμε στην οργάνωση των επιχειρήσεων κάτι το οποίο μπορεί να ενισχύσει τη θετική εικόνα της Ευρώπης, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι πάρα πολύ καλή αυτή η εικόνα. Πιστεύουν ότι η Ευρώπη απλώς ε, κάνει υπερβολικές ρυθμίσεις, αλλά δεν βοηθά τις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λεγκρίπ. Ευχαριστώ κύριε ε, Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, θα ήθελα να ανοίξω λίγο το... Ε, να διευρύνω το φάσμα της συζήτησής μας, να σας ρωτήσω ε, τι σας λέει ο μεγάλος πρωταθλητής ε, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και αν πιστεύετε ο μεγάλος πρωταθλητής ε, είναι ο ανταγωνισμός, αυτός είναι πραγματικά που δημιουργεί μεγαλύτερη επιχειρηματικότητα. Ξέρω ότι δεν είστε απολύτως υπεύθυνος γι' αυτό και αρμόδιος γι' αυτό, αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι στο κομμάτι που σας αναλογεί, ε, θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Κύριε Επίτροπε. Ε, ε, Ευχαριστώ. Απαντάω κατευθείαν στην κυρία Βάιλερ για την που πρέπει να ευχαριστήσω για την πολύτιμη δουλειά τη και για τα όσα έκανε με την οδηγία για τι καθυστερήσει πληρωμών. Η υποχρέωσή μου είναι να γίνει σεβαστή σε όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μικρέ, μεσαίε, Μεγαλύτερε άσχετα και με την πολιτική απόχρωση τη κυβέρνηση Είναι ηθική η υποχρέωση. Πληρωμές πρέπει να γίνονται στις επιχειρήσεις, γιατί οι επιχειρήσεις, εφόσον συνεργάζονται με το δημόσιο, πρέπει να πληρώνονται. Κινδυνεύουμε σε αυτή την περίοδο της κρίσης να πεθάνουν λόγω έλλειψης πιστώσεων οι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα λοιπόν ε, ε, ξανά και ξανά στη διάρκεια τη συζήτηση αυτή. Θα έρθω σε επαφή με όλε τι κυβερνήσει, ακόμη και με αυτέ που ακόμη δεν έχουν μεταφέρει την οδηγία ή δεν έχουν κοινοποιήσει αυτό, δεν το έχουν κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Γερμανία δεν την έχει μεταφέρει την πρόταση οδηγία. Η Γαλλία. Η Γαλλία έχει ορίσει ένα χρονοδιάγραμμα, αλλά ελπίζουμε να το ακολουθήσει. Δεν θέλω τώρα να μπω σε μια τέτοια κουβέντα για τα εσωτερικά τη ομοσπονδιακή δημοκρατία τη Γερμανία, Αλλά καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και κόντρες μεταξύ των κομμάτων, όμως υπάρχουν και δυσκολίες γραφειοκρατικές. Κάποιοι προτιμούν τι δημοσιονομικές πολιτικές και σε αυτές δίνουν έμφαση αντί στι αναπτυξιακές. Και στην ε, χώρα μου, τη χώρα καταγωγή μου, πρέπει να πληρώνονται, πρέπει να πληρωθούν πολλά οφειλόμενα ποσά ακόμα και αναδρομικά. Καταλαβαίνω λοιπόν τη δυσκολία, όμως θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να επαγρυπνούν για να γίνει σεβαστή πλήρωση η οδηγία. Θα έρθω σε επαφή με τα δύο αρμόδια υπουργεία στην Γερμανία για να λάβω τις απαραίτητες πληροφορίες και να σας δώσω τις απαραίτητες διευκρινήσεις για την μεταφορά. Εάν χρειαστεί η Γερμανία κάτι επιπλέον σε ό,τι αφορά την εναρμόνιση των φορτιστών. Όπως είπα πριν από λίγες μέρες λάβαμε επιστολή από πλευράς οκτώ παραγωγών. Μετά την απόφασή μου να προχωρήσουμε ενεργότερα αποφάσισαν να δηλώσουν προθυμία να αναλυθεί η πρωτοβουλία. Αναλύουμε λοιπόν από τεχνικής πλευράς την επιστολή. Εάν η πρωτοβουλία μου Κάπω πιεστική οδηγήσει σε εθελοντική επίλυση του προβλήματος, ευχαρίστω. Θα σταματήσω κι εγώ το αμάξι μου και την όλη ατμομηχανία αυτή τη πρωτοβουλία και θα επιτρέψουν να συναυθεί συμφωνία μεταξύ των παραγωγών. Αυτή θα ήταν η ιδανική κατεύθυνση. Όμω και το κείμενο που εσεί ετοιμάζετε προ τη σωστή κατεύθυνση οδηγεί. Διότι επιτρέπει να δοθούν συγκεκριμένε λύσει για του πολίτε. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση τη κυρία Καρνιέτη. Η ανάπτυξη συνεχίζει να είναι προτεραιότητά μας. Στις 17 και 18 Ιουνίου για την Ρώσια θα είμαστε στην Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη. Μετά τον Ιούλιο θα ο Επίτροπος Ποτότσνικ με ε, αντιπροσωπεία εκπροσώπων της πράσινης βιομηχανίας θα είναι στην Κίνα. Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές Σκοπεύουμε να πάμε στη Μιανμάρ, στο Βιετνάμ και μέσα, μέχρι το τέλος του 2014 στον Καναδά και την Αυστραλία. Βέβαια, μετά θα πρέπει να ρωτήσετε τον επόμενο επίτροπο εάν σκοπεύει να ολοκληρώσει το γύρο αυτών των επισκέψεων. Πάντω, η δική μου Γενική Διεύθυνση και οι συνεργάτε μου ευχαρίστω να σα δώσουν όλε τι απαραίτητε πληροφορίε για επιχειρήσει που σκοπεύουμε να επισκεφθούμε και για να δηλώσετε συμμετοχή εφόσον θέλετε σε οποιαδήποτε από αυτέ τι πρωτοβουλίε. Τα δημοσιεύουμε και στον ιστότοπό μα, αλλά αν θέλετε να έρθετε σε επαφή με τι υπηρεσίε και να ενημερώνεστε τακτικά για αυτέ τι πρωτοβουλίε, ευχαρίστω. Και όσο αφορά την ερώτηση τη κυρία Λεγκρίπ, ήδη συζητούμε ως Ευρωπαίοι σε διεθνέ επίπεδο. Υπάρχουν κανόνες της που πρέπει να γίνονται σεβαστοί. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε ή αν έχουμε την ευκαιρία να αναθεωρήσουμε τους κανόνες για τις κρατικές ε, βοήθειες που ο κύριος Αλμούνια μόλις ε, υπέβαλε σχετική πρόταση στο Σώμα των Επιτρόπων, στο Συλλογικό Σώμα για τον αντίκτυπο του ανταγωνισμού και για την προάσπιση, την προστασία της ανταγωνιστικότητας. Έχουμε τους κανόνες του 1957, όπου η ανταγωνιστικότητα και ο ανταγωνισμός μεταξύ Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Βελγίου ήταν κάτι που περιοριζόταν στις χώρες αυτές. Σήμερα ο διεθνής ανταγωνισμός είναι κάτι που πρέπει να μας ε, απασχολήσει Πώς θα επιτρέψουμε στι ευρωπαϊκές επιχειρήσει να αναμετρηθούν με κινέζικες, ινδικές, ρωσικές, αμερικανικές, βραζιλιάνικες. Πρέπει να το σκεφτούμε το θέμα. Ναι, δεν είναι ταμπού. Εγώ διηγούμε πάντοτε μια σύντομη ιστορία. Το πρώτο μου μάθημα ως φοιτητή δικαίου στο Πανεπιστήμιο, ο καθηγητής φιλοσοφίας του δικαίου μας ρώτησε «Ξέρετε γιατί το δικαστήριο χτίστηκε δίπλα στο ποτάμι και απάντησε γιατί το δίκαιο δεν αλλάζει. Ο νόμος είναι αυτός που μεταβάλλεται προκειμένου να εφαρμόζεται σωστά το δίκαιο. Η ανταγωνιστικότητα λοιπόν είναι μια κινητήριος δύναμη για να ενισχυθεί η οικονομία την αφαρμογή των νόμων όμως για την ε, προάσπιση της αξίας της ανταγωνιστικότητας, αυτό είναι κάτι που να το βλέπουμε συχνά. Κατά καιρού, από καιρού καιρό πρέπει κάτι να αλλάζει. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει οι κανόνες ανταγωνιστικότητας να ανοίγουν τις πόρτες σε όλους. Εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πρέπει να υπάρχει και ένα επίπεδο επιπλέον. Κανόνες ανταγωνιστικότητας δηλαδή που επιτρέπουν στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μπορέσουν να αγωνιστούν σε διεθνές επίπεδο. Πρέπει να σκεφτούμε εάν λόγω χάρη μια επιχείρηση κερδίσει ένα διαγωνισμό στην Κίνα και η ευρωπαϊκή επιχείρηση αναγκαστεί να έχει σχέσεις εξωτερικής ανάθεσης και επειδή είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές τους ξεχάσουν όλους και δεν πάρουν καμία ευρωπαϊκή επιχείρηση ως συνεργάτη τι πρέπει να κάνουμε. Νομίζω σε όλους τους τομείς, ας πούμε στη Χαλιβουργία. Και το έχουμε συζητήσει, το έχουμε συζητήσει και με τον κύριο, τον συνάδελφό μου, τον κύριο Έτιγκερ. Έχουμε την ίδια θέση. Πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας προς το εξή. Πού θα παίξουμε παιχνίδι. Πού θα κάνουμε παιχνίδι. Εάν παίζουμε μόνο σε ευρωπαϊκό γήπεδο, είναι διαφορετικό το πράγμα από το αν παίζουμε παγκοσμίω θα υπάρξουν διαφορετικοί κανόνε για τις κρατικές βοήθειες, όπως είπαμε, από τον Επιτροπό Θα τα δούμε, αλλά το Κοινοβούλιο. Εδώ δεν υπάρχει αδιάλακτη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει να συζητήσουμε μεταξύ μα. ναι, ναι. Να δούμε αν υπάρχει λύση. Εάν μας αρέσουν αυτά που γίνονται, όπω σήμερα, κανένα πρόβλημα. Είναι μια θέση. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη την παγκοσμιοποίηση. Δεν υπάρχει Σοβιετική Ένωση. Η Κίνα είναι η Κίνα του σήμερα. Το Μεξικό και η Βραζιλία είναι και άλλε χώρε. Δεν είναι η Βραζιλία του 1957. Η Αφρική. Πώ θα εξελιχθεί τα ερχόμενα χρόνια. Πρέπει όλα αυτά να τα, να τα σκεφτούμε. Διότι αυτό είναι ο ρόλο των πολιτικών ανδρών και γυναικών. Να σκεφτούν και να διαδούν τι θα συμβεί τα ερχόμενα χρόνια. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πάντοτε ότι η πρώτη μα μέρη είναι να προσπιστούμε την αρχή τη ανταγωνιστικότητα, αλλά πώ. Τι πρέπει να κάνουμε. Εγώ λέω ότι κατά πρώτον σίγουρα πρέπει να το συζητήσουμε το θέμα. Ευχαριστώ πολύ ε, που ήρθατε. Νομίζω είχαμε μια πολύ ζωντανή συζήτηση. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε ε, τα θέματα αυτά, τις εποπτείες αγοράς, τα θέματα των ραδιοφώνων και άλλα. Ε, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Για τελευταία φορά στο διαρθωμένο μας διάλογο, είναι ο τελευταίος ετήσιος κύκλος αυτός, θα σας στείλουμε όμως και άλλη πρόσκληση για να επανέλθετε περί το τέλος της θητείας για να κάνουμε μια ανασκόπηση των όσων από κοινού θα έχουμε πετύχει. Ευχαριστώ. Εδώ ολοκληρώνεται η συνεδρίαση της Επιτροπής μας Αμέσως μετά ακολουθεί η συνεδρίαση των συντονιστών. Παρακαλώ όσοι δεν ε, συμμετέχετε στους συντονιστές ε, να ε, φύγετε το συντομότερο από την αίθουσα. Αύριο το πρωί ραντεβού στις 9 με πρώτο θέμα προσβασιμότητα των ιστοτόπων οργανισμών του δημοσίου τομέα. Θα έχουμε και παρουσίαση και στις 10 ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρετε.